Είναι ήδη 3 και 10 και εγώ προτιμώ να είμαι ακριβή. Λοιπόν, αρχίζουμε την απογευματινή μας ακρόαση με θέμα τον εθελοντισμό. Και είναι η πρώτη ακρόαση του νεοεκλεγέντος κοινοβουλίου και αποφασίσαμε να το διοργανώσουμε νωρίς, νωρίς, νωρίς, σήμερα δηλαδή, και δεδομένου το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των κοινωνιών μας, αφορά την εθελοντική προσφορά υπηρεσίας και πολλές φορές υποτιμάται στην Ευρώπη, αντίθετα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ πιστεύω ότι ο εθελοντισμός πρέπει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει πολλές προκλήσεις και γι' αυτό πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερο κύρος σε αυτό το θέμα και πρέπει να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε το 2011 να ονομαστεί έτος του εθελοντισμού και γι' αυτό έχουμε ονομάσει και έναν εισηγητή, τον συνάδελφό μας, ε, Μάρκος Κούρια, ο οποίος ε, είναι και ο εισηγητής της ε, γνωμοδότησης και θέλουμε την έκθεση αυτή να την ολοκληρώσουμε ε, υπό σουηδική έκθεση αυτή να την ολοκληρώσουμε προεδρία. Έχουμε επίσης ε, μέλος του, του πάνελ, τον κύριο Παύλο Τζουζέπε, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ένωσης Εθελοντικών Οργανισμών, τον ε, κύριο Πίτερ ε, Williams, ο οποίος είναι πρόεδρος της, του οργανισμού Adult Resources και του προσκοπικού οργανισμού της προσκοπικής κίνησης στο Βέλγιο, ε, τον ε, Δόκτωρ Πάολο Τζουζέπε Ντικάρ, Γενικό Διευθυντή της Ιταλικής ε, Υπηρεσίας Εθνικής Νεότητας Ιταλίας και έναν δικό μας συμπατριώτη, ο οποίος είναι Διευθυντής των Εθνικών Οργανώσεων στο Βέλγιο, τον κύριο Μάρκους Χέλτ. Νομίζω κατάγεται από το Βερολίνο, αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ θα μιλήσει εκ του Βελγίου. Έχουμε επίση επίσης τον φίλο μας Πιέρ Μερέστα, και τον κύριο Ένρικ Σέλιν από την ε, τότε, Βρετανική ε, περίοδο της Προεδρίας, διότι είχαμε συζητήσει το θέμα τότε επί Βρετανικής Προεδρίας. Είχαμε αποφασίσει να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη και να το ολοκληρώσουμε. Αυτή η ακρόαση είναι δημοφιλής, όπως βλέπετε έχουμε και πολλούς επισκέπτες και θα συζητήσουμε εθελοντικές δράσεις, προγράμματα και θέλουμε να προβάλλουμε περισσότερο τις εργασίες που κάνουν αυτά τα εθελοντικά στελέχη αλλά και το έργο των οργανώσεων ε, οποίες, ή για τις οποίες εργάζονται. Καταρχάς θα γίνει μια γενική παρουσίαση και συζήτηση για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη και εν συνεχεία θα απαντήσουμε στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο για την στήριξη του εθελοντισμού. Εάν θέλουμε το 2011 να γιορτάσουμε τον εθελοντισμό πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η προστιθέμενη αξία του εθελοντισμού στην Ευρώπη και τι πρωτοβουλίες πρέπει να αναλάβουμε ε. που θα συμβάλλουν σε αυτή την προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω δίνοντας το λόγο καταρχάς στον εισηγητή, τον κύριο Μάρκο Σκούρια, ο είναι εισηγητής της νομοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερος ε, σημαντική γιατί έχουμε σήμερα την δυνατότητα να ακούσουμε ε, Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες ε, για το θέμα αυτό και ε, ένα θέμα ε, στο οποίο πραγματικά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πρέπει να μετρηθούμε σαν Ευρώπη, γιατί ο εθελοντισμός είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα μάλα της ε, κοινωνίας μας να προοδεύσουν, αλλά να βελτιώσει και τον κάθε ένα πολίτη να βελτιωθεί προσωπικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε σήμερα εδώ εκπροσώπους σωματείων, οργανισμών, οργανώσεων και τοπικών ε, οργανώσεων. Δεν, ε, δεν θα ήθελα να κλέψω ε, υπερβολικά πολύ χρόνο από τους ομιλητές. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω εάν πραγματικά πρέπει τώρα να αναφερθώ στην ε, έκθεσή μου ή μήπως να δώσουμε πρώτα τον λόγο στους προσκεκλημένους μας και μετά να ολοκληρώσουμε με τη δική μου παρέμβαση. Επομένως, ε, σας ξαναδίνω τον λόγο. Εντάξει, τότε να δώσω το λόγο στον, ε, στον δόκτωρο Ντικάρο να κάνει εκείνο την εισήγησή του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το Προεδρείο της Επιτροπής, ε, τον εισηγητή, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας εδώ πρέπει να εκφράσω την μέγιστη ικανοποίησή μου για την προσοχή με την οποία φαίνεται να παρακολουθεί το Κοινοβούλιο το θέμα του εθελοντισμού ε, και το οποίο σχετίζεται και με άλλα ζητήματα τα οποία όπως είπε και ο εισηγητής κ. Σκούρια πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της ευρωπαϊκής διαδρομής, έτσι ώστε να βελτιωθεί όχι μονάχα η σχέση της Ευρώπης με τους πολίτες της, αλλά ε, για να βελτιωθεί η ίδια η Ευρώπη, ε, έτσι ώστε να συντονιστούν καλύτερα τα κράτη και οι κυβερνήσεις αρέσκομαι στο να ξεκινώ με κάποιες ε, γενικές ε, θεωρήσεις. Εγώ βρίσκομαι εδώ κυρίως ε, ως διευθυντής, γενικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Νεότητος της Ιταλίας και σαν εκπρόσωπος του προγράμματος Νεολαία σε δράση. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν ασχολούνται μονάχα οι νέοι με τον εθελοντισμό, Ας το θέσουμε διαφορετικά. Οι νέοι βεβαίως είναι η κινητήρια δύναμη των διαδικασιών αυτών και των διεργασιών ε, που προωθούν την Ευρώπη και επομένως οπωσδήποτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το μέλλον της Ευρώπης. Όμως θα πρέπει να δούμε τον εθελοντισμό στο σύνολό του γιατί ε, βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούμε και την σταδιακή γύρανση του πληθυσμού, ε, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει αφενός να πάρουμε διαφορετικές στρατηγικές από ό,τι στο παρελθόν, ε, και αφετέρου να κάνουμε διαφορετικού είδους παρεμβάσεις πλέον. Έλεγα προηγουμένως ότι ασχολούμε κυρίως με τον αθλητισμό στους ε, νέους και με την νεολαία ε, και βεβαίως ε, βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα όπως είναι τα προβλήματα, τα προσκόμματα μάλλον της κινητικότητας, της διασυνοριακής επαφής και από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσω. Θα πρέπει να ληφθούν ε, τα μέτρα αυτά τα οποία θα διευκολύνουν ε, ακόμα περισσότερο την διασυνοριακή κινητικότητα των νέων. Μια διασυνοριακή κινητικότητα η οποία έχει ήδη ε, ξεκινήσει να γίνεται πραγματικότητα λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που όμως δυστυχώς ακόμα αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Κυρίως δε όταν πρόκειται να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή νέοι ε, που ξεκινούν με συγκριτικά μειονεκτήματα. Επομένως αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, δηλαδή να δούμε τις δυσκολίες των νέων. Έστω και αν σε σχέση με κάποια χρόνια πριν είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κανείς από τη μία χώρα στην άλλη, ακόμα οι νέοι, κυρίως αυτοί που έχουν μικρότερες, λιγότερες δυνατότητες και ευκαιρίες, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνησή τους. Οι πληροφορίες επίσης ε, οι οποίες ε, λαμβάνουν ε, οι νέοι και αντίστοιχα οι πληροφορίες που οι νέοι μπορεί και πρέπει να στέλνουν σε αυτούς που παίρνουν τελικά τις αποφάσεις. Αυτή η κίνηση, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι εύκολη. Τρίτο σημείο είναι το γεγονός του πολλαπλασιασμού των ευκαιριών ε, και η κατάρτιση καταλόγων κατά κάποιο τρόπο με τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί στην Ευρώπη ε, υπάρχουν εξαιρετικές εμπειρίες εθελοντισμού και νεανικού εθελοντισμού ιδιαίτερος. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και λιγότερο νέοι, οι οποίοι έχουν σαν στόχο ζωής ε, τον εθελοντισμό. και πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια του προγράμματος Νεολαία σε δράση αγγίξαμε από κοντά αυτήν την ε, πραγματικότητα ε, και δυστυχώς αντιμετωπίσαμε ε, το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης πόρων και της έλλειψης πληροφοριών που έχουν να αντιμετωπίσουν συχνά οι νέοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τον, ε, ε, με τον εθελοντισμό. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολλοί οι νέοι αυτοί οι οποίοι ζητούν ε, να ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού, αλλά δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα ή λείπουν οι απαραίτητοι πόροι. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ υπερβολικά με το θέμα των ε, πόρων, γιατί ξέρετε όλοι το λένε αυτό και σε πολλές ε, περιπτώσεις. Όμως, όμως, και εδώ επαναλαμβάνω και μία ε, άποψη η οποία είναι ευρύτερα διαδεδομένη στον χώρο του εθελοντισμού, και που είναι αδιαμφισβήτητη. Δηλαδή ότι εάν η Ευρώπη θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της σε ισχυρές γερές βάσεις, θα πρέπει να ε, δώσει πόρους διαφορετικούς και άλλους σε τομείς, που, σε τομείς με τους οποίους ασχολούνται αυθόρμητα εκατοντάδες και ε, χιλιάδες άνθρωποι που το κάνουν αυθόρμητα, που το κάνουν από την καρδιά τους ε, και που δυστυχώς αντιμετωπίζουν έλλειψη πόρων και τρόπων ε, για να παρέμβουν. Πρέπει λοιπόν η παρέμβαση να είναι διαρθρωτική Ζητούμε επομένως διαφορετικές παρεμβάσεις. Ζητούμε οι πόροι να ε, μην αφορούν μονάχα ε, αυτά καθεαυτά τα προγράμματα εθελοντισμού, αλλά να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να βελτιώσουν τη δομή του εθελοντισμού στην Ευρώπη. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο βεβαίω είναι σημαντικό και το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι αυτό της, των, της πληροφόρησης ε, και της ε, ικανότητας να δημιουργηθεί ένα, ε, μια διαδικασία πολλαπλασιαστική. Σήμερα, πέρα από την οποιαδήποτε καλή βούληση ή καλή θέληση των οργανώσεων, πέρα από τα προγράμματα και τα, τα εργαλεία τα οποία ε, βρίσκονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Και δεν είναι πάντα εύκολο να έρθουν ε, οι οργανώσεις σε επαφή με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Πρέπει επομένως οι οργανώσεις, ε, οι διάφορες τα διάφορα σωματεία, τα διάφορα ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με τον εθελοντισμό, να είναι σε θέση να συνδιαλέγονται με αυτούς που ε, παίρνουν τις αποφάσεις. Θα πρέπει να δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις να είναι σε θέση να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Θα πρέπει να ε, θεσμοθετηθούν κάποια ποιοτικά πρότυπα, κάποια ποιοτικά στάνταρ, ε, επί των οποίων θα μπορούσαμε ε, να βασιστούμε, δηλαδή να υπάρχουν ενιαία και ομοιόμορφα ε, στοιχεία ε, βάσει των οποίων να επιλέγονται ε, τα σωματεία ή οι θελοντικές δράσεις. Θα πρέπει επίσης οι οργανώσεις να κατανοήσουν ότι για να μπορέσει κανείς να παρέμβει με ορθό τρόπο θα πρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής τι είδους παρεμβάσεις θα γίνουν, ποια θα είναι η στάση όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις απέναντι στον εθελοντή, απέναντι στην εθελοντική οργάνωση, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε ο εθελοντής να μπορέσει να προχωρήσει σωστά στο δρόμο τον οποίο έχει χαράξει. Πολύ δουλειά μας περιμένει. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ε, η πιστοποίηση. Υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο και αυτό ε, παρεμβαίνει κυρίως όσον αφορά τον εθελοντισμό των νέων. Είναι το Youth Pass. Είναι όμως ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει πλέον να αγκαλιάσει όλες τις μορφές του εθελοντισμού και που θα πρέπει να εναρμονιστεί και αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια, αλλά θα πρέπει λέγω να εναρμονιστεί ε, και με την νομοθεσία των διαφόρων κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής αναγνωρισιμότητα του έργου των εθελοντών. Δηλαδή, ε, θα πρέπει ε, η εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει ο εθελοντής ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιστοποιείται έτσι ώστε να μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιηθεί στην αγορά εργασίας. Αυτό μας το ζητούν οι εθελοντές. Γιατί ξέρετε πολύ συχνά εθελοντικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες που μπορεί να μην είναι μια πραγματική κανονική μαθητεία, αλλά τελικά μπορεί να είναι ένα μεγάλο μάθημα και ένα μεγάλο, ε, ε, μια μεγάλη αποσκευή για τους ε, εθελοντές, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και μάλιστα με τρόπο ίσο και ισοδίκαιο για όλους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν εμπειρίες οι οποίες δεν είναι τυπικές ε, και οι οποίες αφορούν την ίδια την εθελοντική δράση αλλά και την κατάρτιση ε, των εθελοντών ε, είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και ξέρετε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για τους νέους αφού έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όσα έχουν μάθει στη διάρκεια είτε της μαθητείας τους είτε του ίδιου του εθελοντισμού να μην μπορούν λέγω να τα χρησιμοποιήσουν μετά στην επαγγελματική τους ζωή. Τέλος, ε, υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ε, ε, όσον, και, και κατάρτισης και σε επίπεδο οικογένειας και σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, σε επίπεδο σχολείου και επομένως και τα ίδια τα κράτη σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε αποκεντρωμένο επίπεδο θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ένα άλλο επιμέρους θέμα είναι οι εθελοντές με αναπηρία. Υπάρχουν ήδη ευρωπαϊκά προγράμματα ε, τα οποία πραγματικά δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ε, ε, αναπηρία. Δηλαδή οι εθελοντές δεν θα πρέπει ε, διορθώνω, τα άτομα με αναπηρία δεν θα πρέπει να είναι μονάχα αποδέκτες και να θεωρούνται ε, δεδομένα ως αποδέκτες του εθελοντισμού. Θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι σε θέση να προσφέρουν εθελοντική ε, εργασία. Και επομένως η οποιαδήποτε παρέμβαση θα γίνεται, είτε με ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε με άλλου είδους προγράμματα, κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να είναι προσεκτικά Μίλησαμε επανειλημμένα ε, για αυτήν την πύλη, ευρωπαϊκή πύλη των νέων, αυτό το πόρταλ, στο, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο οι νέοι μπορούν να βρουν ε, πολλά στοιχεία. Στο εσωτερικό αυτής της τράπεζας δεδομένων μπορεί μελλοντικά να γίνει η συνολική τράπεζα δεδομένων του εθελοντισμού που προσανατολίζει τους νέους προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει να ενταχθούν ε, μεθοδολογίες, τυπολογίες, ε, γεωγραφική μορφή του, του εθελοντισμού, ιδιαίτερες μορφές, ιδιαίτερες παρουσίες του εθελοντισμού σε διάφορα σημεία και χώρες της Ευρώπης. Όλα τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε αυτήν την πύλη έτσι ώστε όποιος εθελοντής θέλει να ασχοληθεί ε, με κάποια εθελοντική εμπειρία, να μπορεί να το κάνει και εάν κάποιος εθελοντής θέλει ο ίδιος να δημιουργήσει ε, μια νέα εμπειρία δική του, να μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από αυτό το πόρταλ, από αυτή την πύλη. Στο δεύτερο τμήμα της παρέμβασής μου θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, προτάσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι προσπαθώντας να εστιάσουμε την προσοχή στα προβλήματα ε, διαφαίνονται άμεσα και οι πιθανές και δυνατές λύσεις και επομένως η καθημερινότητά μας μας φέρνει αντιμέτωπους αφενός με τα προβλήματα αλλά και αφετέρου και ταυτόχρονα με τις πιθανές λύσεις. Θα σταματήσω εδώ επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγή προσανατολισμού ε, στον εθελοντισμό και αρχίζω, τελειώνω συγγνώμη από εκεί που ξεκίνησα. Δεν μας ενδιαφέρουν ε, κάποιες ε, τομεακές συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μας ενδιαφέρει μια συνέχεια και μια συνέπεια όσον αφορά τον εθελοντισμό όσον αφορά τους εθελοντές, σε αυτούς που κάποια στιγμή της ζωής τους αποφασίζουν να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή και να αφιερωθούν στην κοινωνία. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους ε, η προσοχή θα πρέπει να είναι δεδομένη, ε, προσοχή λοιπόν στους εθελοντές, ε, στον εθελοντισμό, στην κινητικότητα των νέων κυρίως, προσοχή απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να βασιστεί σε πολύ γερές βάσεις. Σε μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να έχει πολυπολιτισμική ε, προσέγγιση και που θα βασίζεται στην αμοιβαία γνωριμία. Γιατί μονάχα εάν γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, μονάχα εάν τα μέλη της ε, κοινότητας ε, γνωρίσουν οι μεν τους δε, μονάχα τότε λέγω θα, μπορεί, θα μπορέσει να υπάρξει η πραγματική ενσωμάτωση. Ε, διαφορετικές παρεμβάσεις ε, λοιπόν όσον αφορά τον εθελοντισμό και θα ασχοληθώ με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις και τις πιθανές ε, δυνατές λύσεις, πιθανές δυνατές πρωτοβουλίες. Με αυτές θα ασχοληθώ στο δεύτερο τμήμα της παρεμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λαντσάνο τώρα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω το εξής. Με εμφανίζεται ως ε, ε η υπεύθυνο του ΣΠΕΣ του Κέντρου Στήριξης των Εθελοντών της Ρώμης, αλλά ε, είμαι και υπεύθυνο ε, για, για την ευρωπαϊκή διάσταση του εθελοντισμού. Και ε, το τονίζω αυτό γιατί δεν θέλω η παρέμβασή μου να είναι εθνοκεντρική, να είναι εθνική. Θα ήθελα αντιθέτως να επιστήσω την προσοχή όλων ημών στην ε, εργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντισμού γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην κοιτάμε μονάχα τη δικιά μας χώρα ή τη δικιά μας πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδιαλεγόμαστε ε, με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αλλά και με ε, την Ευρώπη μέσω των θεσμικών της οργάνων. Είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω σε αυτήν την ε, συνάντηση, αλλά δεν με τελικά, γιατί παρακολουθώ την προσπάθεια του Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια ε, όσον αφορά τον εθελοντισμό και πρέπει να πω ότι πραγματικά το Κοινοβούλιο έχει συμβάλει τα α, μάλα ε, και στο θέμα του εθελοντισμού, αλλά και στο να ε, θεσμοθετηθεί το έτος 2011 ως, ως έτος του εθελοντισμού και οπωσδήποτε καθορίζονται ε, κάποια πολύ σταθερά στοιχεία τα οποία θα μας ε, ε, βοηθήσουν και στην σημερινή μας συζήτηση. Δηλαδή να δούμε πού και πώς πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και το 2011 αλλά και από τώρα μέχρι το 2011. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί ξέρετε δεν με την πυρίτιδα σήμερα Απλώς σήμερα βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτόν τον μακρύ δρόμο του εθελοντισμού. Ε, ε, του εθελοντισμού που ε, από ένα παραμελημένο θέμα τελικά έχει βγει στο προσκήνιο και καλεί την προσοχή των πολιτών αλλά και των κυβερνήσεων και των κρατών. Να σας πω λοιπόν εξ αρχής ότι σήμερα δεν υπάρχει και αυτό το βλέπουμε και στο, ε, στη δυσκολία του να βρούμε το πραγματικά σωστό όνομα ε, για το ευρωπαϊκό έτος. Δεν υφίσταται, λέγω σήμερα, ένας ορισμός για τον ε, ευρωπαϊκό εθελοντισμό. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύση ακριβώς μέσω των πρωτοβουλειών ε, που θα ε, κινητοποιήσουμε για το 2011 και μέχρι το 2011. Ε, θα πρέπει το, ο εθελοντισμός να έχει κοινά στοιχεία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και εδώ υπάρχει κάποια δυσκολία. Γιατί υπάρχει μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά την, τοποθέτηση της ε, κοινωνίας ε, των ε, πολιτών απέναντι στον εθελοντισμό. Βλέπουμε δηλαδή και σε σχέση με το 2011 συμμετέχουν ας πούμε οργανώσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να οριστούν σαν εθελοντικές οργανώσεις, σαν οργανώσεις εθελοντισμού μάλλον. Αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεπεράσουμε. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν υπάρχουν στατιστικές ε, με τις οποίες ε, να συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχουν καν στατιστικές, γιατί η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ε, δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Και επομένως, εάν θέλουμε να στηρίξουμε με κάποιο τρόπο την δράση των εθελοντών και τον εθελοντισμό, θα πρέπει να αναλύσουμε ε, αυτήν την δράση, να δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι εθελοντές, με ποιο τρόπο κινούνται, μέσω ποιων οργανώσεων, με ποιο τρόπο κτλ. Και αυτό θα πρέπει να το λύσουμε μέχρι το 2011. Το επόμενο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το εξή. Από πολιτική απόψεω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, δεν έχουμε ακόμα σαφή αναγνώριση των ε, ε, υπηρεσιών είτε ε, σε επίπεδο μεμονωμένων κυβερνήσεων είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε σαφή αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχουν οι εθελοντές και οι υπηρεσίες εθελοντισμού. Και ε, τόσο στις τομεακές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο ε, και στις ε, πολιτικές των μεμονωμένων κρατών μελών ο εθελοντισμός παραμένει ένα από τα τελευταία στοιχεία σε καμία περίπτωση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και ίσως μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζεται οργανικά κατά κάποιο τρόπο η σημασία, η, αυτοτελής λοιπόν σημασία το, του εθελοντισμού. Ε, στην ε, χώρα μου υπάρχουν ε, διάφοροι νόμοι, οι οποίοι όμως δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τον εθελοντισμό και επομένως θα πρέπει να αναλυθεί με μια μεγάλη πολιτιστική πρωτοβουλία έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών, το κομμάτι της τουλάχιστον που ασχολείται με τον εθελοντισμό θα πρέπει να αναγνωριστεί και να θεσμοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως ε, υπάρχει και μία σειρά ειδικών ε, στοιχείων τα οποία δεν ε, αναγνωρίζονται. Ας πούμε ο προλαλής σας αναφέρθηκε στην μη αναγνώριση προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης και που δεν αναγνωρίζονται λοιπόν ως τυπικά προσόντα. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσουμε και κατά αυτή την έννοια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον εθελοντισμό σαν ένα ε, εκ των βασικών συστατικών της ε, ε, σύγχρονης δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Για να περάσουμε σε πιο απλά καθημερινά ζητήματα, να πω το εξής. Λυπούμεθα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δείχνει να συντονίζεται ε, στις διάφορες υπηρεσίες της ε, οι οποίες ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να συνδιαλεγόμαστε εμείς σαν εκπρόσωποι του εθελοντισμού με ε, κάποια υπηρεσία της Επιτροπής. Δεν υπάρχει λοιπόν ενιαία αντιπροσώπευση είτε από την πλευρά τη Επιτροπή είτε από την πλευρά των εθελοντικών οργανώσεων. Επομένω, θα πρέπει ε, να βρεθεί καλύτερο τρόπο ε, συντονισμού. Έστω ε, ακόμα και όταν συζητάτε η χρηματοδότηση των διαφόρων πρωτοβουλειών και μέσα στα πλαίσια των δράσεων που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάχυση ε, που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Θα θέλαμε λοιπόν ε, να ε, έχουμε έναν συγκεκριμένο συνομιλητή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα μας βοηθούσε και θα μας βοηθούσε επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα ότι το, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στηρίξει τον εθελοντισμό, θέλει να στηρίξει τα ευρωπαϊκά δίκτυα εθελοντών. Επίσης, ε, ε, βλέπουμε ότι μέχρι τώρα τα προγράμματα στήριξη του εθελοντισμού είναι βραχυπρόθεσμα, είναι ενός ε, δύο ετών. Εμείς θα θέλαμε μια, μια, μια πιο μακρόπνοη πολιτική. Θα θέλαμε επίσης διαρθρωτική χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων με τρόπο ώστε να μην δίνεται δημόσιο χρήμα χωρίς να ξέρουμε ακριβώς σε ποιον το δίνουμε και για ποιο λόγο ε, θα θέλαμε να θέσουμε τον εθελοντισμό σε πολύ σαφείς και γερές βάσεις και επομένως ε, και εμείς να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρει πού δίνει τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ε, ovviamente non è direttamente collegata al 2011 ma σε σχέση με το 2011 θα ήθελα να φέρω ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν αφορά μονάχα το 2011 δεν υπάρχει ενιαία νομική βάση για τον εθελοντισμό. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ειδικό νομικό πλαίσιο, άλλες χώρες στις οποίες και αυτό απουσιάζει, δεν υπάρχει καθόλου δηλαδή νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν. Ε, σε, σε ορισμένες χώρες με, με, με μεγάλη εμπειρία στα κοινωνικά ε, θέματα ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η έλλειψη, το πρόβλημα αυτό τη έλλειψη τη νομική βάση έχει λυθεί κατά το μάλλον ή τον ικανοποιητικά. Όμω στι νέε χώρε ε, το πρόβλημα παραμένει έντονο. Στι νέε αυτέ χώρε, ε, εννοώ τι χώρε οι οποίε πρόσφατα έγιναν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όπου η κοινωνία των πολιτών ακόμα είναι λίγο μετέωρη όσον αφορά ε, την δυνατότητα οικοδόμησης ε, κοινών, ε, κοινωνικών αγαθών. Εκεί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, τίθεται διαρκώς και επομένως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να λυθεί. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα πλαίσιο αναφοράς έστω για αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζουν τον εθελοντισμό και επομένως να οριστούν κάποιοι πυλώνες επί των οποίων να στηριχτεί η ε, κοινωνική δράση και η εθελοντική δράση στις ε, χώρες ε, αυτές. Ας πούμε, στις χώρες αγγλοσαξονικής παράδοσης τα πράγματα ε, έχουν λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες ε, στις οποίες ακόμα η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Θα σας δώσω τώρα και κάποιο παράδειγμα. Η ασφάλιση των εθελοντών. Δεν συζητιέται το θέμα αυτό, ούτε καλύπτεται νομικά σε όλες τις χώρες. Όμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για εθελοντές, ε, μιλάμε για δραστηριότητες οι οποίες ε, ακριβώς προσφέρονται εθελοντικά. Το να χρεωθεί ο εθελοντής με τα έξοδα της ασφάλισης του, ε, πραγματικά αυτό αποτελεί τροχοπέδι ε, και παρεμπόδισε κατά κάποιο τρόπο της εθελοντικής δραστηριότητας. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει κάποια ομοιογενής απάντηση. Δεύτερον, μια εγγύηση ε, κατά το μάλλον ή των ευρωπαϊκού επίπεδου ε, σχετικά με τον εθελοντή, ο οποίος είναι και εργαζόμενος και ο οποίος θα πρέπει να καλύπτεται ε, για τις μέρες για τις οποίες, τις οποίες αφιερώνει στην, στον εθελοντισμό. Θα πρέπει να εγγυηθούμε στους εθελοντές, τους νέους και λιγότερο νέους, την δυνατότητα ε, να ασχολούνται με τις εθελοντικές τους δραστηριότητες. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι οι χρηματοδοτήσεις μέσω των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τον εθελοντισμό, η πρόσβαση ε, σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γιατί ε, τη στιγμή που οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί περίπου σε όλους, δηλαδή και σε εταιρείες και σε επιχειρήσεις ε, και σε ε, διαφόρων μορφών νομικά πρόσωπα και σε εθελοντικές οργανώσεις ε, και όσον αφορά τις δραστηριότητες συγχρηματοδότησης και όσον αφορά την διαχείριση των προγραμμάτων, πρέπει να σας πω ότι ε, οι εθελοντικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά αυτή την έννοια, οι οποίες ε, τις περισσότερες φορές ε, είναι αξεπέραστες. Και υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα ότι με τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται οι διαγωνισμοί και μπορώ κατά αυτήν την έννοια να σας δώσω πάρα πολλά προγράμματα είναι σαφές ότι αυτός ο οποίος προκυρίζει στον διαγωνισμό δεν γνωρίζει καθόλου, μα καθόλου σας διαβεβαιώ, την πραγματικότητα του εθελοντισμού. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί διαγωνισμοί για τους εθελοντές και για τις εθελοντικές οργανώσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαγωνισμών. Ε, ειδικοί διαγωνισμοί λοιπόν που θα επιτρέπουν σε αυτές τις οργανώσεις οι οποίες ε, πραγματικά προσφέρουν ε, εξαιρετικό έργο, γιατί έχει υπολογιστεί ότι το 5% του ΑΕΠ ε, βασίζεται στην εθελοντική, παράγεται μάλλον βάσει εθελοντικής εργασίας. Και θα δίνεται επομένως η δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν ο μηχανισμός αυτών των διαγωνισμών να επανεξεταστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ' επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσει την ε, φορολογική, το φορολογικό καθεστώς των εθελοντικών οργανώσεων, είτε με μείωση, αν όχι, ε, ε, αν όχι ακύρωση του ΦΠΑ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθελοντικοί οργανισμοί προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες, δεν πληρώνονται με κανένα τρόπο για τις υπηρεσίες ε, οι οποίες, ε, ε, οι οποίες προσφέρονται και επομένως δεν είναι δυνατόν μετά να φορολογούνται με 25% για τις υπηρεσίες αυτές που δωρεάν έχουν προσφέρει. Δύο πραγματάκια ακόμα και τελειώνω. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ούτε εθνικές πολιτικές υπάρχουν, στήριξη της αναδιάρθρωσης του εθελοντισμού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ε, ως ε, ε, οργάνωση συζητήσαμε και την τελευταία, στην τελευταία μας συνάντηση στην Σουηδία. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ουσιώδες ζήτημα εάν θέλουμε ο εθελοντισμός να αναπτύξει το δυναμικό του και τις δυνατότητές του. Ο εθελοντισμός ε, σε πολλές χώρες και σε πολλές περιπτώσεις ε, γίνεται ε, μέσα από οργανώσεις των 10 ατόμων με προϋπολογισμό που δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ το χρόνο. Ε, και παρόλα αυτά αυτού του είδους ο εθελοντισμός δίνει τρομερά αποτελέσματα. Συμμετέχει στο, στο ΑΕΠ, συμμετέχει στην μαθητεία, στην εκπαίδευση. Επομένως, ο, η αναδιάρθρωση η οποία σημαίνει βοήθεια και στήριξη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες υπάρχει εθελοντισμός χωρίς όμως ταυτοχρόνως να υπάρχει η δομή που θα στηρίξει τον ε, ε, εθελοντισμό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταίο κάτι που είπε και ο συνάδελφος Δικάρο. Θα πρέπει να ε, δυναμώσουμε χρηματοδοτώντας τις και περισσότερο τις πολιτικές ε, ανταλλαγών, τις πρωτοβουλίες ανταλλαγών. Προγράμματα ανταλλαγών που δεν θα αφορούν όμως μονάχα τους νέους. Βεβαίως θα πρέπει να αυξηθούν τα προγράμματα αυτά για τους νέους, αλλά όχι μόνο για τους νέους. Εμείς στη δικιά μου οργάνωση Μόλις ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε σύντομα στις ε, Βρυξέλλες, ε, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών ε, ηλικιωμένων ατόμων, συνταξιούχων. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Ενίας ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαπιστώνοντας την επιτυχία ε, του προγράμματος αυτού είναι διατεθειμένη να δώσει ακόμα περισσότερες χρηματοδοτήσεις, συλλαμβάνοντας δε υπόψη ότι το 2012 θα είναι μάλλον το έτος συνεννόησης μεταξύ των ηλικιών. Επομένως θα πρέπει ε, πραγματικά να ε, δοθούν περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια έτσι ώστε οι ανταλλαγές να είναι περισσότερες και να χρηματοδοτούνται καλύτερα. Ε, θα πρέπει να ενδυναμωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία, η διεργασία των ανταλλαγών, γιατί είναι ένα στίχημα για το μέλλον. Ευχαριστώ. thank Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρατσάνο και συνεχίζουμε με τον κύριο Πίτερ Βίλεμς και μετά θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε. Θα προσπαθήσω ε, να παρουσιάσω την ε, ομιλία μου αυτή. Χτες το βράδυ είχα δύο συναντήσεις, το βράδυ, οπότε κανονικά πρέπει να πάρω άδεια για σήμερα. Είναι πάντα δύσκολο να οργανώσει κανείς μέσα σε λίγο χρόνο τέτοιες παρουσιάσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας μιλήσω λοιπόν για τις θελοντικές οργανώσεις. Οργανώσει, ή για οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν με θελοντές. Οι θελοντικές οργανώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την ε, πολιτική που ακολουθούν ανάλογα με το αν έχουν πληρωμένο προσωπικό, διοικητικό προσωπικό επίσης. Και σε τι διάρκεια χρόνου απασχολούν εθελοντές. Θα αναπτύξω τέσσερα σημεία. Μερικά έχουν ήδη υποθεί έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα τα πω κι εγώ. Εξάλλου είπαμε, εθελοντές δεν πληρώνονται. Πρώτον, αυτό που μας χρειάζεται είναι αναγνώριση, να μας αναγνωρίζει η κοινωνία. Ορισμένοι νομίζουν ότι οι πρόσκοποι που για παράδειγμα δραστηριοποιούνται πολύ στην ε, Φλάνδρα και στην Ευρώπη γενικότερα κάνουμε babysitting. Και ότι πληρωνόμαστε. Όχι. Εμείς αυτό που παίρνουμε σαν αμοιβή είναι η προσφορά μας στην κοινωνία. Η νομοθεσία, αν αλλάξει επίσης, μπορεί να βοηθήσει να διευκολύνει τη ζωή των εθελοντών και των προσκόπων, αλλά και άλλων εθελοντικών οργανώσεων που δεν έχουν πλαίσιο. Αυτό όμως που βοηθάει είναι την ανάπτυξη του ατόμου ο Και αυτό βέβαια με έναν τρόπο άτυπο. Και αυτό πρέπει να παραμείνει, να είναι άτυπος. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η έλλειψη χρόνου που, έχουν, ε, που υπάρχει σήμερα για τους εθελοντές. Γιατί οι εθελοντές συνήθως είναι μαθητές ή σπουδαστές και δεν έχουν χρόνο για να προσφέρουν έργο στην κοινωνία. Άσε που υπάρχει και κάποιο αίσθημα ανταγωνισμού Πώς παραμένει μια οργάνωση εθελοντική ελκυστική απέναντι σε μια άλλη. Έπειτα υπάρχουν όλο και νέα συστήματα για project. Και χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να καταφέρει κανείς να βρει το δρόμο του μέσα σε αυτά. Και πολλές φορές λέει άσε. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η έλλειψη κινήτρου. οι νέοι δεν θέλουν τη σημερινή ημέρα να ασχολούνται με διοικητικό έργο, να κάθονται σε ένα γραφείο. Θεωρούν ότι είναι όλο αυτό πολύ γραφειοκρατικά και ότι δεν μπορούν να προσφέρουν καλό έργο έτσι. Γι' αυτό η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί. Γιατί τελικά Πολλέ φορέ δεν καταφέρνουμε καν να δαπανίσουμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε. Κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με τα κίνητρα των εθελοντών είναι ότι ένας εθελοντής αναρωτιέται πολλές φορές γιατί να φάω το χρόνο μου όταν έχει την αίσθηση ότι δεν προσφέρει κάτι επικοδομητικό, αλλά απλώ κάθεται πίσω από ένα γραφείο. Έπειτα, το τέταρτο σημείο μου είναι οι πόροι. Ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι που διατίθεται. Έτσι κι αλλιώς ένα project κοστίζει πολύ σε χρόνο. Λείπει ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά οι εθελοντές. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. So, thank you very much for your ευχαριστώ πολύ. picture. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Έχουμε τώρα μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων, των προβλημάτων και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση έτσι ώστε τα μέλη της Επιτροπής μας να αποτανθούν προς το πάνελ αν έχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Yes, please. Merci, madame. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάτι για την ορολογία. Ξέρω μερικές φορές ότι η ουσία και ο τύπος ε, παίζουν ρόλο. Εδώ μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και αλλού της εθελοντικής προσφοράς. Αυτά τα δύο όμως δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ο εθελοντισμός σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταμοιβή είτε οικονομική είτε άλλη. Οπότε, για να μπορεί κανείς να καταλάβει καλύτερα και πιο σωστά, θα ήθελα να αλλάξουμε το κείμενο και να μιλάμε για το ευρωπαϊκό έτος της προσφοράς εθελοντικής εργασίας και όχι του εθελοντισμού. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο αυτό. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα υπάρχει μόνο στα γαλλικά, λέει ο Μιλήτρια. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Βίλεμς που αναφέρθηκε στους προσκόπους. Εγώ συμμετέχω σε μια ένωση ε, ατόμων που είναι γονείς προσκόπων. Η η ιδέα αυτή της προσφοράς χρόνου, της έλλειψης αμοιβή είναι πράγματα τα οποία για τους νέους μας σημαίνει μεν όχι αμοιβή, σημαίνει όμως ανάληψη ευθύνη. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί όταν είμαστε 18-20 ετών, αν έχουμε την ευθύνη για 10-12 παιδιά, δεν είναι κάτι απλό. Ούτε για έναν ενήλικα, πόσο μάλλον για έναν νέο 18. Ευχαριστώ. Ωραία. Να ακούσουμε μερικέ ερωτήσει. Σχόλη κυρία Κώστα. Ε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, τις ε, εισηγήσει αυτές γιατί μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία εκκίνησης όπως άλλωστε και η έκθεση του εισηγητή μας. Να θέσω κάποια ερωτήματα. Πρώτον, γίνεται μία προσπάθεια αλλαγής του ονόματος του έτους, ε, έτσι ώστε να γίνει ευρωπαϊκό έτος, όχι εθελοντισμού, αλλά εθελοντικών δράσεων. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, μάλλον όχι, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι από τη μία μεριά έχουμε τις ανάγκες της επικουρικότητας, ε, την, ε, την πλευρά δηλαδή και της του πλούτου που έχει κάθε χώρα αφενός ε, και, και των ιδιαιτεροτήτων που έχει ε, κάθε χώρα, αλλά από την άλλη πλευρά ε, του γενικότερου πλαισίου που θα πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο έτσι ώστε οι εμπειρίες να είναι συγκρίσιμες και έτσι ώστε ο εθελοντισμός να είναι σαν αντίληψη ίδιος σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, ε, τι θα πρέπει να έχει, ποια στοιχεία θα πρέπει να διαθέτει, ποια χαρακτηριστικά μία ε, οργάνωση έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί ε, στην, στο έτος αυτό ή στις δραστηριότητες που αναγνωρίζουμε εμείς ως εθελοντικές. Και νομίζω ότι είναι σαφές ε, σε όλους μας ε, ότι για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόθεση η διάθεση να ε, ε, προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν πραγματικό συντονισμό ε, των εθελοντικών δράσεων. Δηλαδή, ναι, να αναλυθούν πρωτοβουλίες στη διάρκεια και στα πλαίσια του έτους, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση για κάτι παραπάνω. Τρίτον, όταν λέτε, αναφέρεστε σε δίκτυα νέων, ε, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στα δίκτυα που έχουν ε, εθελοντική ε, μορφή. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς συντονίζονται τα δίκτυα αυτά μεταξύ τους και με τι ακριβώς ασχολούνται. Και επίσης θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας σχετικά ε, με ε, τις επενδύσεις που θέλετε να γίνουν στο μέλλον ε, σχετικά με το πώς θέλετε να κινηθείτε. Επίσης, τρίτη ηλικία. Εμείς πάντα σκεφτόμαστε την τρίτη, τα άτομα της τρίτης ηλικίας σαν αποδέκτες των εθελοντικών δράσεων και όχι σαν εθελοντές. Ε, νομίζω ότι είναι αλήθεια λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο ε, τα θέματα αυτά γιατί άλλωστε η δημογραφική πορεία της ε, Ευρώπης ε, είναι ε, δεδομένη και επομένως κατά αυτή την άποψη θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα σε αυτή την ομάδα στόχο να δώσουμε λίγο περαιτέρω και επιπλέον δυνατότητες να τους δώσουμε τη δυνατότητα να φέρονται σαν να είναι ακόμα νέοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τίκης. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ε, ακροατές που ήρθαν σήμερα το απόγευμα. Είναι μια, ένα σημαντικό ζήτημα ο εθελοντισμός ή η προσφορά εθελοντικής εργασίας μου επιτρέπετε ως μέλος μιας ε, ε, ε, χώρας της Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης να μιλήσω από την οπτική γωνιά ε, του δικαίου των δικαιωμάτων των πολιτών κάτω από ένα δικτατορικό καθεστώς υπό τις συνθήκες αυτές ε, τα προσωπικά, οι προσωπικές ε, δυνατότητες, ε, τα προσωπικά αιτήματα είχαν καταπιεστεί, εκμηδενιστεί και το άτομο είχε ισοπεδωθεί. Οι ελευθερίες αυτές αποτελούν, οι ανύπαρτες αυτές ελευθερίες θα αποτελούσαν τη βάση των εθελοντικών δράσεων. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντική η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην Ευρώπη για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και εθελοντικές υπηρεσίες, η προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ε, ο ρόλος των εκκλησιών είναι επίσης πολύ σημαντικό όταν, σημαντικός, όταν το 1998 ε, δόθηκε πολιτική, ε, θρησκευτική ελευθερία και μπορέσαμε να ανοίξουμε τις εκκλησίες, πάρα πολλές εκκλησιαστικές οργανώσεις ανέλαβαν εθελοντικές ε, δράσεις. Μέχρι τότε οι ενέργειες αυτές ήταν απογορευμένες, δεδομένου ότι οι εκκλησιαστικές και θρησκευτικές δραστηριότητες απαγορεύονταν υπό το καθεστώς. Η διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών θα γίνει σύντομα και ο πρόεδρος κύριος Χούζακ θα υποδεχθεί μία αντιπροσωπεία ε, των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων εκκλησιών. Ένας διάλογος εξαιρετικά χρήσιμος. Με αυτή τη συμπλήρωση λοιπόν του σκέλους, του στοιχείου της συμβολής των εκκλησιών, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να παρέμβω. Ο κύριος Σκέλη. Ευχαριστώ. Οι ομιλητές μας ε, έδωσαν μια θαυμάσια εικόνα, μια γενική εικόνα του εθελοντισμού και της ε, έλλειψης αναγνώρισης σε πολλές περιπτώσεις, ε, το οποίο είναι δυστυχώς πολύ λυπηρό. Όλα αυτά, όλες αυτές τις προκλήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν είναι σωστό να είμαστε υπερβολικά αρνητικοί. Βεβαίως, ο τίτλος του πρώτου πάνελ είναι ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθελοντές και αθελοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Εάν δείτε τον αριθμό των εθελοντών στην Ευρώπη, το θέμα της αναγνώρισης της αξίας τους δεν είναι και τόσο σκοτεινό, δεν είναι τόσο αρνητικό. Έχουμε υπολογίσει ότι τρεις από τους δέκα ενήλικες συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα εθελοντική προσδίδοντας αξία με την εργασία τους αυτή, με την προσφορά τους αυτή στην κοινωνία. Βεβαίως, η πρόκληση για μας είναι ότι οι 7 από τους 10 που δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή έχουν πει ότι θα ήθελαν, θα το επιθυμούσαν, αλλά υπάρχουν προσκόμματα που τους εμποδίζουν. Ε, αυτή ακριβώς λοιπόν τώρα είναι η πρόκλησή μας. Εάν το ονομάσουμε το 2011 έτος του θελοντισμού, θα πρέπει τους, ε, οι, οι 7 που δεν συμμετέχουν να τους προσεγγίσουν οι τρεις εθελοντές που συμμετέχουν και να τους πείσουν και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτά τα προσκόμματα που δεν τους επιτρέπουν τη συμμετοχή. Όταν εμείς ε, εκτελούσαμε ορισμένες ε, δράσεις στην Ιρλανδία με τον πρώην Πρωθυπουργό, με την ενίσχυση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Μπέρτι Αχέρν, είχαμε σημειώσει ότι οι άνεργοι και οι ηλικιωμένοι, η τρίτη γενιά δηλαδή, είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες λόγω διαθέσιμου χρόνου να ασχοληθούν με θελοντικές εργασίες. Βεβαίως, ε, το να είσαι άνεργος ε, ε, είναι μία αντίφαση και να προσφέρεις θελοντικά την εργασία σου. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. επίσης, η τρίτη ηλικία, πολλές φορές χρόνο, έχουν και οι εργαζόμενοι που παίρνουν προώρη σύνταξη. Έχουν χρόνο στη διάθεσή τους. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε οι τρεις εθελοντές να αγκαλιάσουν και τους υπόλοιπους 7. Η, τα εμπόδια πρέπει να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν. Ευχαριστώ λοιπόν τους ομιλητές και ε, ψάχνοντας τις λύσεις πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη γενική εικόνα, το ευρύτερο πλαίσιο. Ο εθελοντισμός είναι μάλλον η μία δραστηριότητα η οποία διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα όσο καμία άλλη, διότι η κάλυψη των βασικών αναγκών, ύπνος, φαΐ, στέγαση, είναι, καλύπτονται και από τον άνθρωπο και από τα ζώα. Αλλά ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο <laughs> δεν είναι ούτε ένστικτο, ούτε βασική ανάγκη. Είναι μία προσφορά η οποία γίνεται με μία προσωπική δέσμευση. δέσμευση. λοιπόν ότι το 2011 θα μας δώσει μία θαυμάσια ευκαιρία τους τρεις ε, εκ των 10 να τους κάνουμε 10 εκ των 10, 100% δηλαδή συμμετοχή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη διευκρίνηση, λέει η πρόεδρο, τι ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Και προχωράμε. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες του πάνελ που μου φανήκαν πάρα πολύ ικανοί αλλά και πολύ δεσμευμένοι του εθελοντισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι χαρακτηριστικό για τους εθελοντές. Έρχομαι και εγώ από μια τέως κομμουνιστική χώρα και πρέπει να σας πω ότι το εθελοντικό κίνημα αλλάζει την πραγματικότητα στην Πολωνία. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό κίνημα εθελοντισμού και συμφωνώ μαζί σας κύριε, ξέρω πολλά για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη και στην Πολωνία και θέλω λοιπόν μια σκέψη μου να μοιραστώ μαζί σας. Το κίνημα εθελοντισμού έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο εξαιτίας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εθελοντές και που αντικαθιστούν πολλές φορές τις τοπικές κοινότητες ή ακόμα και την κυβέρνηση σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά είναι τόσο πολύτιμη η εθελοντική αυτή δράση γιατί οι θελοντές είναι και αυτοί πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είναι πολύτιμοι για μας. Σε μια δημοκρατία, σε μια ανοιχτή Ευρώπη, αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές διαδικασίες με αυτόν τον τρόπο, οπότε ανοίγονται στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτόν τον κοινό τόπο και για άλλους. σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τον άλλον. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο μπορεί κανείς να καταλήξει βάσει των εθελοντών που γνωρίζουμε, οι οποίοι δρούν σε διάφορα προγράμματα στην Ευρώπη και είναι οι καλύτεροι Ευρωπαίοι που μπορούμε να φανταστούμε. Αναφερθήκατε επίσης στις εκκλησίες. Τέσσερα χρόνια δούλεψα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήμουνα εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία. Αναφερθήκατε επίσης σε διαγωνισμούς για κάλυψη προμηθειών. Εγώ θυμάμαι ότι μου βάζανε προϋποθέσεις που με εμπόδιζαν να συνεργαστώ με θελοντές. Αυτό είναι πολύ αρνητικό γιατί έτσι, για παράδειγμα, μέναν απ' έξω κάποιες εκκλησίες, κάποιες θρησκευτικέ κοινότητες σε ορισμένε χώρες και αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει την κάθε χώρα να την εξετάζουμε διαφορετικά. Δεν είναι δυνατόν τους εθελοντές να τους βάζουμε ως PR. Εγώ χρειάστηκε να δουλέψω με τέτοιες οργανώσεις και πολύ συχνά θα είχα προτιμήσει να δουλέψω με μη κερδοφόρες οργανώσεις, αλλά δεν μπορούσα εξαιτίας της νομοθεσίας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μας επιτρέπει όταν πρόκειται σε διαγωνισμούς να μπορούν να συμμετάσχουν και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης πρέπει να γνωστοποιήσουμε το κίνημα εθελοντισμού. Όπως γίνεται με το Εράσμους Μόντους ή με το Σόκρατς. Πρέπει να το κάνουμε και για τον εθελοντισμό αυτό. Ε, Ευχαριστώ θερμά. Ich τους ε, ομιλητές. Πριν ξεκινήσουμε είχα κάτσει λίγο να σκεφτώ τι σημαίνει αυτό το έτος 2011 ε, ε, και τέσσερα σημεία εντόπισα, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Καταρχάς, τι εικόνα παρουσιάζει ο εθελοντισμός και η εθελοντική εργασία δεν είναι πια η εικόνα των ανθρώπων που έχουν σκύψει από το βάρος της εργασίας και των ετών, αλλά είναι άνθρωποι με ε, δράση, με δύναμη, είτε είναι νέοι είτε είναι πιο ηλικιωμένοι, που πράττουν, ενεργούν συνειδητά και θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πού μπορούμε να ε, εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους στη διαβίου μάθηση και σε άλλες εθελοντικά προγράμματα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μία ε, εικόνα της κατάστασης στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν θέλουμε τα πάντα βεβαίως να γίνουν και να αποφασίζονται στην, ε, στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και τις τοπικές αρχές. Όπως ξέρετε, εθελοντισμός ε, σημαίνει έξοδα, παρόλο που είναι εθελοντισμός. Ε, καταρχάς, εκπαίδευση, ε, κατάρτιση, αποστολή κάπου, να δουλέψεις εθελοντικά. Βεβαίως, ε, ανταμείβες 100% με το προσφερόμενο έργο, αλλά πολλές φορές χρειάζεται συντονισμός να, να παρουσια... και επίσης ε, μοντέλα τα οποία πρέπει να παρουσιάσεις, να στείλεις δηλαδή προσωπικό να παρουσιάσει ή να εκπαιδεύσει. Άρα λοιπόν ο θελοντισμός δεν είναι όλα δωρεάν και τζάμπα, ε, υπάρχουν και έξοδα που πρέπει να γίνουν. Τρίτον, Υπάρχουν πολλές φορές φόβοι και επιφυλάξεις ότι δεν θέλουν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν εθελοντές διότι φοβούνται ότι δεν θα κάνουν καλά τη δουλειά τους επειδή δεν πληρώνονται. Ενώ εγώ πιστεύω ότι αυτός που έχει μέσα του το, το κύτταρο του εθελοντισμού είναι αυτός που είναι και περισσότερο δεσμευμένος. Και τέταρτον, ίσως αυτό είναι χαρακτηριστικό γερμανικό πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κανένας δεν έχει το φόβο ότι η εθελοντική εργασία ακυρώνει τις ε, θέσεις εργασίες που πληρώνονται. Δηλαδή ότι θα χάσουν κάποια άνθρωποι τη δουλειά τους επειδή ορισμένοι θα έρθουν εθελοντές και θα πάρουν τις θέσεις τους. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η φοβία πολλοί συνεργάτες μας, οι οποίοι ήταν μισθωτοί, είχαν αυτό το φόβο, ε, αυτό τον ενδόμηχο φόβο, ο, τι θα γίνει τώρα που πρέπει να κάνουμε οικονομίες, μπας και καταργήσουν τις θέσεις μας και φέρουν εσελοντές να δουλέψουν στα, στην καρέκλα μας. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Ο κύριος Τάκουλα, κυρία Μπέρντερ μετά. Δεν έχουμε και πολύ καιρό. Σύντομα παρακαλώ. Um, σας ευχαριστώ. Και εγώ έρχομαι από τον τομέα του εθελοντισμού και έχω δουλέψει για χρόνια εκεί. Χαίρομαι ειλικρινά πολύ για το όσα ακούμε για τον εθελοντισμό. Βλέπετε, είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου να μαζευτούν το έτος εθελοντισμού και να ανταλλάξουν τις καλύτερες πρακτικές και τις εμπειρίες τους γενικότερα είναι πολύ σημαντικό, είτε πρόκειται για ανθρώπους που βοηθάνε στα νοσοκομεία, όπω ακούσαμε σε εκκλησίες ή αλλού. Εγώ δούλευα ε, για... και βοηθούσα ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε δύσκολη κατάσταση στην κοινωνία. Όλοι όσοι έχουν δουλέψει στον αθελοντισμό ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες, ξέρουν ότι χρειάζονται στήριξη είτε πρόκειται για κατάρτιση, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Όπως επίσης αναγνώριση. Όταν αφήσουν τη δουλειά τους στην εθελοντική, να μπορούν να αποδείξουν εκεί που θα πάνε να ζητήσουν δουλειά, τι έκαναν τον καιρό που ασχολιόντουσαν με τον εθελοντισμό. Πολλοί που δούλεψαν στον εθελοντισμό έφυγαν αναγνωρίζοντας ότι έχουν κερδίσει πάρα πολλά από την περίοδο του εθελοντισμού από την περίοδο της προσφοράς τους. Κάποιος πριν αναφέρθηκε στον εφιάλτη της χρηματοδότησης και είναι εφιάλτης για μας. Αν μπορούμε λοιπόν με το έτος αυτό βοηθήσουμε να αφαιρεθεί ο ΦΠΑ, ήδη αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά για τους εθελοντές. Έπειτα το να βρει κανείς τη χρηματοδότηση όντω είναι δύσκολο γιατί πρέπει να βρεις αυτό που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες και είναι ένας εφιάλτης ειλικρινά. Θα έπρεπε και αυτό να το δούμε το έτος εθελοντισμού. Έπειτα, να μοιραστούμε καλύτερα τη γνώση μεταξύ μας. Κάποιες χώρες δεν έχουν αυτό, ε, αυτή την παράδοση. Εγώ έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και για μας το Ηνωμένο Βασίλειο η παράδοση είναι τεράστια στον εθελοντισμό. Έχουμε πραγματογνωμοσύνη, ξέρουμε εμπειρίες, οπότε ας περάσουμε αυτή την εμπειρία και σε άλλους. Δηλαδή ε, κατά τη διάρκεια του έτους εθελοντισμού ας φροντίσουμε να περάσουμε τη γνώση και την εμπειρία μας σε αυτούς που δεν την έχουν. Αν το πετύχουμε αυτό, το έτος εθελοντισμού θα στεφθεί από επιτυχία. Ο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ και εγώ σε αυτό το θέμα που πιστεύω ότι είναι πραγματικά εξαίρετο. Υπάρχουν πολλές μορφές έκφρασης εθελοντισμού. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, έχουμε πάνω από 6.000 εθελοντές και είναι κάτι που εκτιμά όλος ιδιαίτερος. Ακούσαμε ότι το έτος 2011 θα είναι το έτος εθελοντισμού. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην ηθική αξία του εθελοντισμού. Πρόκειται για ηθικές αρχές οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή. πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο επιλέγονται οι εθελοντές για να κάνουν ποια δουλειά, κατά πόσο οι εθελοντές όντως χρησιμοποιούνται για τη δουλειά εκείνη την οποία γνωρίζουν καλύτερα. Οι περισσότεροι εθελοντές είναι νέοι, αυτό είναι καλό. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι μετά από ένα διάστημα στη φυλακή θέλησαν να μπουν στην εθελοντική εργασία. Είτε πρόκειται για ανθρώπους που καταδικάστηκαν για παιδεραστή, είτε άλλους. Όπως και να έχει πάντα το πράγμα, αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι ενδιαφέρον είναι να προχωρήσουμε προσεκτικά και να φροντίσουμε οι χώρες μας να συμμετέχουν στον εθελοντισμό για όποιου είδου οργάνωση και αν πρόκειται. Πιστεύω πάντως ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή που πήραμε. Κύριε Πακ, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στη γλώσσα μου, στα ρωματικά δηλαδή. Έκανε χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα έχω διανύσει. Με συνοδεύει ραβίνος από το Ισραήλ και θέλω να θίξω ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν ξέρω κατά πόσο αύριο θα μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσω. Έχω μόνο ένα-δύο λεπτά στην αυριανή μου παρέμβαση. Πάντως, είμαι κοινωνιολόγος με δεκτορικό στην, ε, στις θρησκείες και θέλω να προτείνω στην Επιτροπή μας να φτιάξουμε μία υποεπιτροπή για να προστατεύσουμε τα ιερά κημητήρια, τις εκκλησίες της Ευρώπης, διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με εβραϊκά ε, νεκροταφεία στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου, διακόπτη πρόεδρος. Αγαπητέ μου κύριε Μπάντεμ, εδώ έχουμε μία ακρόαση με θέμα τον εθελοντισμό <coughs> δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συζητάμε, συζητάμε εδώ πολλά προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει. Αλλά σήμερα μιλάμε στα πλαίσια μιας συγκεκριμένη ακρόση επί ενό συγκεκριμένου θέματος. Και το θέμα αυτό, εθελοντισμός, το συζητάμε. Εάν δεν θέλετε να παρέμβετε με, με κάτι σχετικό, παρακαλώ να μιλήσετε την επόμενη φορά υπό το σημείο διάφορα. Πολύ λυπάμαι, αλλά εδώ υπάρχουν κανόνες και πρέπει να, τις, να τους στηρίσουμε. Η κυρία Μακλά. Next time in committee. Την επόμενη φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όποτε θέλετε μπορείτε να μιλήσετε ε, για το δικό σας θέμα. Σήμερα όμως έχουμε καλέσει ομιλητές Ωραία, αύριο μου επιτρέπετε. Δύο λεπτά. Ναι, αλλά εγώ είμαι μέλος, ε, λέει στην κυρία Πακ, ε, όπως και εσείς. Εντάξει, ελάτε αύριο, λέει η κυρία Πακ, αλλά αύριο δεν θα είναι κανείς εδώ, γιατί δεν έχουμε συνεδρίαση. Η κυρία Μακάρθη έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τόσα όσα μας είπατε. Εδώ ο ελεύθερος χρόνος που δίνουν εθελοντέ είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη σήμερα. Συμφωνώ μαζί σας πάντως ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, η οποία εμποδίζει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό. Αλλά βλέπετε πολλά πράγματα δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές. Η συμμετοχή στον εθελοντισμό εμποδίζεται από το κόστος και τη γραφειοκρατία. Αυτά τα δύο λοιπόν πρέπει να αφαιρεθούν. Αλλιώ, νομίζω ότι θα υπήρχαν πολύ λιγότερα προβλήματα. Έπειτα η αναγνώριση που λέτε των ε, εθελοντικών οργανώσεων όντω είναι και αυτή σημαντική. Και αυτό ακριβώ κάνουμε εδώ σήμερα. Χρησιμοποιούμε τη συνεδρίαση αυτή για να πούμε ότι αναγνωρίζουμε εθελοντικέ οργανώσει, ότι είναι πολύτιμε. Εποφελούμε λοιπόν από αυτή την ευκαιρία για να σας πω ευχαριστώ και να σας πω πόσο πολύ εκτιμάμε την προσωπική προσφορά του κάθε θελοντή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιάκη, είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κι εγώ ε, αγωνίζομαι σε συλλόγους και είχα την ευκαιρία μάλιστα 10 χρόνια να ασχολούμαι στη γαλλική κυβέρνηση με αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν εδώ να αναφερθώ και εγώ σε αυτή τη διαφορά του εθελοντισμού και της ε, εθελοντικής εργασίας. Βολονταριά και μπενεβολά. Ο εθελοντισμός είναι κάτι ιδιαίτερο στη Γαλλία και δημιουργούνται παρεξηγήσεις που δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται. Πολύ. Ε, λοιπόν από εσά που εκφράσετε στα αγγλικά, α κάνετε αυτή τη διάκριση παρακαλώ. Λοιπόν, χαίρομαι και εγώ που έχουμε αυτό το έτος και με εκπλήσει που βλέπω πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Οι οργανώσεις διαφέρουν μεταξύ τους, ο τρόπος που ασκείται η θελοντική εργασία είναι πολύ διαφορετικός Φυσικά έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια στο κίνημα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τους εθελοντές ή τις εθελοντικές δομές, αυτές είναι οι μη κερδοσκοπικές και είναι κάτι άλλο, μην τα μπερδεύουμε όλα, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί, μην γενικεύουμε και μην προσπαθούμε με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλους όσους ανήκουν σε αυτή την ομάδα, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφοροποίησεις. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι στην Ευρώπη εμείς ζητάμε συνεχώς από τις αθλητικές οργανώσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στις κοινωνίες μας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και να επιμείνουμε να υπάρξει και μία πολιτική διάσταση. Εγώ άκουσα τον κύριο Τάκουλα και συμφωνώ μαζί του όταν μιλάει για την ηθική διάσταση που πρέπει να τη δούμε. Όντως, υπάρχει το θέμα της ηθικής, υπάρχει το, πράγμα και το θέμα της δημόσιας τάξης, αλλά προσοχή, δεν μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε όλον αυτό το πλούσιο κόσμο, ας αφήσουμε τον κάθε πολίτη να οργανωθεί όπως επιθυμεί. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάικιν, μια που είναι η συγγήτρια. Ε. Παρακαλώ, κυρία Χάικιν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ναι, όντω έφτασα αργά και ζητώ συγγνώμη, ήμουν σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Ξέρετε ότι για να πάει κανεί από τη μια άκρη στην άλλη του κοινοβουλίου, το σπαθάμε σύντομη. Δεν άκουσα τη συζήτηση, αλλά όπω και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι και εγώ Χαίρομαι πάρα πολύ που το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Αθελοντισμού. Την τελευταία φορά είχαμε γραπτή δήλωση στο προηγούμενο κοινοβούλιο δηλαδή και η επιθυμία μας έγινε πραγματικότητα. Χαίρομαι γι' αυτό. Μία παρατήρηση μόνο έχω να κάνω γιατί άλλα σίγουρα έχουν υποθεί. Σίγουρα θα αναγνωρίσουμε την αξία της θελοντικής εργασίας. Επίσης, πολλές θελοντικές οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη περιμένουν από εμά να κάνουμε κάτι στην πράξη. Και αναγνωρίζω, ναι, ότι το θέμα ε, του να πούμε πόσο πολύ αναγνωρίζουμε την εθελοντική εργασία και λοιπόν όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά να πάρουμε και μια πρωτοβουλία και θα σα δώσω εδώ ένα παράδειγμα που νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποια συνεισφορά εθελοντική σε κάθε ευρωπαϊκό project. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σαν συγχρηματοδότηση. Να λοιπόν κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το προωθήσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Κάτι συγκεκριμένο λοιπόν. Και όλα τα άλλα τα οποία είπαμε βέβαια, δεν λέω σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά να και κάτι πρακτικό που μπορούμε να προσφέρουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα και εγώ έχω να κάνω μερικά σχόλια παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαγωνισμοί διαρθρώνονται με τέτοιο τρόπο όπου εθελοντικές οργανώσεις αποκλείονται. Δεν διαθέτουν τη δομή, δεν διαθέτουν δημόσια κονδύλια. Οπότε, αν εμείς δεν φροντίσουμε να δώσουμε το καθεστώς που τους πρέπει στις εθελοντικές οργανώσεις για να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ε, ποιος θα το κάνει. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και μερικές φορές δεν είναι πολύ πρόθυμη να αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλοί νέοι θέλουν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Και αυτό μέσα από μια θελοντική οργάνωση. Αλλά αυτή η προσφορά πρέπει κάπου να, κάπως να αναγνωρίζεται είτε με ένα Europass είτε όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι πρέπει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν αυτό το έργο στις εθελοντικές οργανώσεις. Αλλιώς θεωρείται σαν χαμένος χρόνος, ενώ δεν είναι, γιατί έχουν αφιερώσει τη δουλειά τους στην κοινωνία και αυτό πρέπει να μπορούν να το αναγνωρίσουν. Θα ήθελα η Κομισιό να προωθήσει περισσότερο μια υπηρεσία τρίτης γενιάς αν θέλετε, senior service. Δηλαδή να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν πάρει σύνταξη και είναι ηλικιωμένοι να είναι δραστήριοι, να μπορούν να προσφέρουν στα καινούργια κράτη, στις νέες δημοκρατίες, στην Αλβανία, στη Βοσνία. Πάντοτε ρωτάω, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί τέτοιες οργανώσεις. Δεν κοστίζουν και πολλά λεφτά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι δύο, αυτές είναι δύο ιδέες που πολύ χρήσιμες και εφικτές. Σχετικά τώρα με το δεύτερο μέρος της ακρόασής μας, προτείνω να κάνουμε το εξής. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, διότι θα πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα. Νομίζω ότι η σύζυγός του είναι ετοιμόγενη και ο νέος μπαμπάς πρέπει να είναι στο πλευρό της. Του εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά και θα του δώσω το λόγο και εν συνεχεία θα ξαναζητήσω από τα μέλη του πάνελ μας να απαντήσουν και να μιλήσουν και για το δεύτερο θέμα, το δεύτερο ερώτημα δηλαδή της ακρόασης. Γιατί και εγώ πρέπει να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα. Έχω να σε μια άλλη συζήτηση. Χαιρόμαστε κύριε Σίλη που μπορείτε να μας διαθέσετε ακόμα λίγο χρόνο αυτή την εξαιρετικά ευτυχή μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ε, όχι, δεν γεννάει αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου. Έχουμε ραντεβού με τον γιατρό. Και όντω κλείνει τους 9 μήνες. Σήμερα. 9 μήνες εγκυμοσύνης. Πράγμα που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή περιμένουμε. Και ίντω ε, να έχουμε ένα νέο εθελοντή σύντομα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, να εκπροσωπήσω δηλαδή την Προεδρία. Ως Πρόεδρος, ε, λοιπόν, της ε, ε, Επιτροπής για Εθελοντικά Θέματα. Ακούσαμε την πρόταση που έγινε τον Ιούνιο. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την άποψή μας όσον αφορά αυτό το θέμα και πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο για να ληφθεί γρήγορα μια απόφαση. Πρώτα απ' όλα όμως, δύο λόγια για να ξεκινήσουμε. Πρώτον, πιστεύω και η Σουηδία πιστεύει ότι κάθε κοινωνία που θέλει να είναι μια λειτουργική δημοκρατία πρέπει να στηρίζει την κοινωνία των πολιτών. Και η κοινωνία των πολιτών, όπως γνωρίζουμε, βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην εθελοντική εργασία. Βέβαια, τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. δούμε όμως τι γίνεται στη δικιά μου χώρα, πάνω από 50% των ανθρώπων στη Σουηδία δίνουν πάνω από 15 ώρες το μήνα σε εθελοντικές δραστηριότητες. Δεν πρόκειται για έναν μικρό τομέα. Πρόκειται, όπως σας είπα, για έναν ακρογωνίο λίθο της δημοκρατίας. Καλύπτει και προσφέρει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και προσφέρει σε όλες τις ηλικιακέ ομάδες της κοινωνίας. Τώρα, πόσο τα κράτη στηρίζουν αυτόν τον τομέα, τι βοήθεια του δίνουν. Αυτό εξαρτάται. Στα κράτη-μέλη δηλαδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η Σουηδία πιστεύει ότι η στήριξη αυτή του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζεται στην έννοια της εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της ακαιρεότητας και της αυτονομίας των εθελοντών. Αυτό είναι κάτι που η Σουηδία θέλει να το υπογραμμίσει, ότι ναι πρέπει να υπάρχουν μέτρα στήριξης, τα μέτρα αυτά στήριξης πρέπει να βασίζονται στην, ε, στο σεβασμό της αυτονομίας του εθελοντή. Εν όψη τώρα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντικής Εργασίας. Είχαμε την πρόταση της Επιτροπής τον Ιούνιο που μας πέρασε. Ξέραμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε έντονες απόψεις για αυτό το θέμα και ότι επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από αυτούς που πρότειναν την οργάνωση αυτού του έτους. Οπότε για μας από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι η υπόθεση αυτή ήταν μια υπόθεση στην οποία θα έπρεπε να αποφασίσει το Συμβούλιο με νομική βάση που απαιτεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε δηλαδή, αν δεν έχουμε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, να πάρουμε κάποια απόφαση. Τον Ιούλιο αρχίσαμε να δουλεύουμε. Το Κοινοβούλιο δεν ήταν ε, διατεθειμένο συζητήσει εκείνη την εποχή γιατί είχε άλλα ζητήματα, οπότε πρέπει να περιμένουμε το νέο Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές δηλαδή, τη σύσταση του σώματος και έτσι συναντηθήκαμε και με τον κύριο Σκούρια, τον εισηγητή, 13 Οκτωβρίου. Τότε είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Παράλληλα με τη δουλειά αυτή, στην ομάδα μου, Επιτροπή Πολιτισμικών Υποθέσεων προχώρησε πολύ. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για κάτι πάνω στο οποίο υπήρχε συνένεση. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε εμπόδια επί της ουσίας. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες από τα κράτη-μέλη. Γενικά η πρόταση της Επιτροπής στηρίχθηκε από τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, ήρθα σε επαφή ίσως όχι με ολόκληρο τον τομέα εθελοντικής εργασίας, αλλά με πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις για να δω ε, την δικιά τους άποψη για την πρόταση. Κάποια από τα θέματα πάνω στα οποία συζητήσαμε και κάποια τέθηκαν και εδώ από ορισμένους πριν, ήταν τα εξή. Κάποιοι είπαν σε ορισμένες χώρες ότι το κείμενο σέβεται την διαφοροποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη πώς δηλαδή οργανώνονται και εκτελούνται οι εθελοντικές εργασίες. Ορισμένες χώρες θέλανε ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην πρόταση να είναι όσο γίνεται περισσότερο ευρύς. Να μην δηλαδή περιορίζει την εθελοντική εργασία έτσι ώστε να αντιστοιχεί ε, στο εργορισμένων οργανώσεων σε ορισμένες χώρες και όχι αλλού. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές εθελοντικής εργασία. Ορισμένες χώρες επίση θέλανε περισσότερες διευκρινήσει για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια κατά το έτος ε, αυτό το Ευρωπαϊκό εθελοντική εργασία. Οπότε, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εθελοντική εργασία, ότι προσφέρει στην οικονομία, στην κοινωνία, πριν όμως από αυτό, Πρόκειται για την ανάπτυξη του ατόμου και για την έκφραση αλληλεγγύης των εθελοντών. Και ορισμένα κράτη-μέλη είπαν ότι αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι αυτό είναι το βασικό. Ότι τα ωφέλη που έρχονται είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να έρθουν σε δεύτερη σειρά. Η σημερινή ακρόαση που οργάνωσε πολύ καλά το Κοινοβούλιο, έχει διάφορα ζητήματα και προβλήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε και το καταλαβαίνετε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού είναι ένα μέτρο για να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θελοντές. Σίγουρα το ευρωπαϊκό αυτό έτος δεν είναι η λύση. Το λέω γιατί όταν τελικά ληφθεί η απόφαση αυτή είναι σημαντικό να ξέρουμε και να ξέρει και ο τομέας τι να περιμένει από αυτό το έτος. Είναι προφανές λοιπόν ότι πολλά προβλήματα πρέπει να λυθούν μακροπρόθεσμα, δεν θα λυθούν όλα μέσα στο ευρωπαϊκό έτος εθελοντικής εργασίας. Αυτό το έτος θα βοηθήσει. Ίσως θα βοηθήσει να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να τα συνειδητοποιήσουμε και μετά να αρχίσουμε να τα λύνουμε. Όπως είπα και πριν, όταν μιλάμε στους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων, είναι ξεκάθαρο ότι παρόλο που υπάρχουν ένα σωρό διαφορές, οι προσδοκίες τους από το έτος αυτό, το ευρωπαϊκό, είναι τεράστιες. Γι' αυτό λέω όταν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό αυτό έτος ότι όλες οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να ξέρουν τι να περιμένουν. Να μην περιμένουν περισσότερα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Στο Συμβούλιο έχουμε σίγουρα μεγάλη φιλοδοξία να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο, να δούμε κατά πόσο μαζί με το Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να υιοθετηθεί η απόφαση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο κύριος Κούριο, ηγητής σας, μας διευκρίνησε και τις δύο φορές που συναντήθηκα μαζί του, ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει όσο γίνεται πιο γρήγορα σε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προκειμένου να καταλήξουμε σε απόφαση όσο γίνεται πιο γρήγορα κι εμείς. Συγχρόνως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να προσπαθήσει να λάβει υπόψη του κάποιες ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωβουλευτές. Δεν είναι βέβαια κάτι εύκολο και έτσι καλώ δεν χρειάζεται συναπόφαση από το Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, η Προεδρία και η ομάδα εργασίας μας ελπίζει και προσδοκά να έχει συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Κι εγώ το ελπίζω αυτό, ότι θα τα καταφέρουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχω πολλές ελπίδες ότι θα πετύχουμε συμφωνία και η απόφαση θα ληφθεί σύντομα. Αυτά προς το παρόν. Τώρα αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Σελήν. Πιστεύω ότι όσοι εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια πρέπει και να ακούγονται όσοι εκλέγονται άμεσα. Όσοι εκλέγονται έμεσα στο πόστο τους, στο Συμβούλιο π.χ. Εύχομαι να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των εισηγητών μας όπως του κυρίου Σκούρια. Γιατί οι προτάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σημαντικά. Εάν θέλουμε το 2011 να το ονομάσουμε έτος του εθελοντισμού, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, στην Κομισιόν. Ο κύριος Μέρες θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εντάξει, δεν είμαι και Θεός. Γρήγορα κάπως θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όλοι συνειδητοποιούμε την ανάγκη που υπάρχει για θελοντική εργασία και για την Επιτροπή. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, στο θέμα τη διάκριση βολονταριά μπενεβολά στα γαλλικά θα επανέλθω αργότερα. Και τα δύο πάντω. Προ το παρόν θέλω να σα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τι κοινωνίε μα. Ξεκινήσαμε από του νέου, είναι αλήθεια. Το ξέρετε όλοι. Ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία η οποία έχει φτιαχτεί με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει μεγάλη επιτυχία, πρέπει να πω. Όλοι οι εθελοντές που συμμετέχουν εκεί είναι περήφανη. Δεν φτάνει όμως. Και συνεχίζουμε. Νομίζω ποιο ήταν ο κύριος Κάρο που είχε πει ότι η μετακίνηση των θελοντών σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί ένα, μια δυσκολία. Πάντως όλες οι χώρες συμφώνησαν να διευκολυνθεί η μετακίνηση αυτή. Αναφερθήκατε επίσης στο Youth Pass, Aeropass Πώς δηλαδή θα αναγνωρίζει κανείς το έργο των εθελοντών και την γνώση που αποκτάνε και την εμπειρία που αποκτάνε από την εθελοντική εργασία. Τώρα σιγά σιγά προχωράμε και επεκτείνουμε τον εθελοντισμό σε όλες τις γενιές. Όσοι είναι δραστήριοι στην αγορά εργασίας ή όσοι βρίσκονται στην ανεργία δυστυχώς και οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, όλοι αυτοί μπορούν να συμμετέχουν. Πριν, ποιο ήταν ο κ. Ροτζάνο, νομίζω, είπε ότι τελικά δεν γνωρίζουμε καλά την κατάσταση όσον αφορά την εθελοντική εργασία στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα. Κάποιο άλλο είπε ότι υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία. Άρα το τοπίο είναι περίπλοκο. Ξεκινήσαμε όμω μία μελέτη και όταν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Έτο Εθελοντισμού θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να μην είναι στατιστικέ τη Eurostat, αλλά θα είναι μια πανευρωπαϊκή μελέτη για τον εθελοντισμό. Έπειτα υπάρχουν διάφορα προγράμματα που σιγά σιγά ενδιαφέρονται και για του λιγότερο νέου εθελοντέ. Να, ο κύριο Τάκουλα ήταν εισηγητή του προγράμματο για του Ευρωπαίου πολίτε ή το Lifelong Learning, κυρία Πρόεδρε το γνωρίζετε πολύ καλά, και αυτό έχει μια διάσταση εθελοντικής εργασίας για τους ηλικιωμένους. Και θα επανέλθω γιατί νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Αλλά ας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Έτος αυτό καθ' αυτό. Πρώτα απ' όλα, πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, ε, στην οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εισακούστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα εγκρίνει τελικά, ελπίζω, το Συμβούλιο. Να λοιπόν, ο καθένα βάζει το πετραδάκι του. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να δουλέψω με τέτοια συμμαχία εθελοντών, γιατί η κοινωνία των πολιτών έχει οργανωθεί. Και να εδώ βλέπω και κάποιους που γνωρίζω και σας το λέω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συνεργάζομαι μαζί σας. Ένα ευρωπαϊκό έτος λοιπόν για κάθε είδους εθελοντική εργασία. Γλωσσικά, ναι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση του νομικού κειμένου, αλλά και στις ανακοινώσεις που θα κάνουμε, στον τρόπο που θα μεταφέρουμε τις προσπάθειές μας προς τα έξω. Δεν πρέπει να αποκλείουμε κανέναν. Είναι πολύ σωστό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν, κάθε θελοντής, ό,τι είδους εθελοντική εργασία και αν προσφέρει. Εξάλλου πιστεύω ότι ο πλούτος, ο μεγαλύτερος πλούτος του ευρωπαϊκού αυτού έτου εθελοντισμού, δεν είναι καν η κοινωνία των πολιτών, παρόλο που είναι πολύ σημαντική. Είναι οι εθελοντέ. Και εγώ θέλω να βρω τρόπο να βάλω μέσα και να συμμετέχουν όλοι οι εθελοντές προσπαθούμε να βρούμε μηχανισμούς μέσω διαδικτύου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να κινητοποιήσουμε όλον αυτό τον πλούτο που είναι οι θελοντές. Ξεκινήσαμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Για παράδειγμα, έχουμε ένα διαγωνισμό για ένα λογότυπο που θα μας προτείνει η κοινωνία των πολιτών. Βέβαια, εννοείται, πρέπει να περιμένω νομικά να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό έτο Εθελοντισμού, αλλά μην νομίζετε ότι περιμένουμε την τελευταία στιγμή για να αρχίσουμε τι προετοιμασίε. έχουμε ήδη αρχίσει. Επίσης, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν κατά το ευρωπαϊκό αυτό έτος εθελοντισμού και οι δικέ μου υπηρεσίες αλλά και των συναδέλφων. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και το είπατε για καλύτερο εσωτερικό συντονισμό μέσα δηλαδή στην Κομισιόν για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό. Είναι κάτι οριζόντιο ο εθελοντισμός και εγώ δεν ε, παριστάνω ότι μπορώ να τα τακτοποιήσω όλα. Έχω συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή άλλους στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν. Όμως ακριβώς αυτό το έτος θα αποτελέσει τον καταλήτη, άμα θέλετε, για να υπάρξει πραγματικό συντονισμός. Για να προχωρήσουμε όμως, το έτος αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να εγκριθεί και αυτό γίνεται πιο γρήγορα ξέρω, κυρία Πρόεδρε, και εσείς και ο κύριος Κούρια, προσπαθείτε και συνεργαζόσαστε με τη Σουηδική Προεδρία για να το πετύχουμε αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στην απόφαση. Πράγματι. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα ευρωπαϊκό έτος δεν οργανώνεται έτσι για πλάκα. Φυσικά και είναι για να προωθήσουμε μια ιδέα, αλλά να ξέρετε ότι απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων, ενέργειας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ε, σταματήσουμε εκεί, πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το ευρωπαϊκό αυτό έτος. Για παράδειγμα, ακριβώς επειδή υπάρχει ποικιλομορφία, υπάρχουν δηλαδή πολλές μορφές εθελοντισμού στην Ευρώπη, το έτος αυτό πρέπει να μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε τις έννοιες να ξέρουμε ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στη συνθήκη δεν νομίζω ότι έχουμε τα μέσα να νομοθετήσουμε. Εξάλλου δεν ξέρω καν αν πρέπει να νομοθετήσουμε για τον αθελοντισμό, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε στις καλύτερες έννοιες, στους καλύτερους ορισμούς της εργασίας αυτής. Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τη διάφορες, πολιτικές. Ο κ. Μπαρόζο πρότεινε ένα πρόγραμμα για το 2020. Όταν θα έχει αποφασίσει για τους επιτρόπους του, θα ξανάρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους επιτρόπους για να προτείνει ένα πρόγραμμα μέχρι το 2015 και ακόμα παραπέρα. Άρα η διάσταση του εθελοντισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη στις διάφορες πολιτικές. Έπειτα, άρση των εμποδίων. Πολλές φορές το ακούσαμε. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να κάνει κάτι, είναι και τα κράτη-μέλη. Μια άλλη τέταρτη πτυχή είναι τα νέα προγράμματα. Γιατί ήδη από τώρα πρέπει να σκεφτούμε τη νέα γενιά ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 31 Δεκεμβρίου 2013 σκεφτείτε ότι είμαστε. Αυτό τι σημαίνει ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει προτάσεις ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο ανάμεση για να εγκρίνουν. Αλλά το 2011 είναι στις πόρτε μας, κοντεύει. Η νέα γενιά λοιπόν προγραμμάτων πρέπει να βάζει μια πιο μεγάλη διάσταση στον εθελοντισμό. Και ίσως, κυρία Πρόεδρε, επί την ευκαιρία αυτή, να διαπιστώσουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μια υπηρεσία εθελοντικής εργασίας των ηλικιωμένων, των seniors. Και τέλος, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού του χρόνου. Πολλά από τα σημεία τα οποία έχουμε ακούσει για την απλοποίηση, η κυρία Χάκιν αναφέρθηκε στην αποδοχή in kind. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για να διευκολύνουμε τη ζωή της, πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή δεν είναι Θεός, είπαμε. Όμως, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό κανονισμό ώστε να έχουν πρόσβαση οι θελοντικές οργανώσεις. Να κάποια στοιχεία που είχα να σας δώσω κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ταπεινοφροσύνη σκέφτεται να βοηθήσει τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Μερές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέλτ που ήρθε λίγο αργότερα επειδή έχει πολλή κίνηση στους δρόμους φαντάζομαι. Έχετε λοιπόν το λόγο και μετά οι εμπειρογνώμονες οι άλλοι. Παρακολουθήσατε ένα μέρος της συζήτησης και πιστεύω ότι έχετε καλυφθεί ήδη σε πολλά σημεία. Πολύ σωστά τα είπετε κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Λέω ο κύριος Χέλτ, με συγχωρείτε γιατί αργοπόρησα. Επιστρέφω από το Βερολίνο στην ίδια πτήση με το Λέχ Βαλένσα και ήμασταν μάρτυρες των, ε, της 20ης επιτίου εχθές στο Βερολίνο από την μέρα που έπεσε το τείχος 11 Νοεμβρίου δεν είναι μόνο τα 20 χρόνια αλλά γιορτάσαμε χτες και την επιτυχία της δέσμευσης των λαών προς την ελευθερία ε, και πιστεύω ότι είναι καλό που σήμερα συζητάμε, τι μπορεί ο κόσμος να προσφέρει, οι πολίτες να προσφέρουν όταν δεσμεύονται για τον εθελοντισμό. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ε, νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε όσον αφορά τον εθελοντισμό. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ε, για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είμαι υπεύθυνο ε, για διάφορε οργανώσει, σαν αυτέ που ανέφερε ο κύριο ε, Μέρε. Ε, αυτή δηλαδή την Ένωση 22 εθελοντικών οργανώσεων. Εγώ όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στις ενδεχόμενες λύσεις. Έχουμε, θα, συμφωνήσω με την, τον εκπρόσωπο της Ειδικής ε, Προεδρίας ε, ότι καλό βεβαίω είναι να έχει κανείς ένα ευρωπαϊκό έτος για τον εθελοντισμό, αλλά είναι πολύ ευρύτερε οι προκλήσεις που έχουμε και τα διακυβεύματα που έχουμε απέναντί μας. Νομίζω, και αυτό μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ κοινότοπο, ε, ε, πιστεύω ότι ο καθένας μας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να είναι εθελοντής. Αλλά ε, όσο κοινότοπο και αν ακούγεται αυτό, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές χώρες στις οποίες και πολλές περιπτώσεις που οι πολίτες δεν μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Ας πούμε, οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε υπηρεσία εθελοντικά. Δεύτερο παράδειγμα. Ε, οι άνεργοι που δέχονται ε, αποζημιώσεις και επιδόματα ανεργίας. Αυτοί δεν μπορούν να προσφέρουν ε, εθελοντική εργασία, γιατί εάν ας πούμε προσφέρουν εθελοντική εργασία για χι ώρες την εβδομάδα ή μάλλον για πάνω από χι ώρες την εβδομάδα, τότε ενδεχομένως θα τους αφαιρεθεί το επίδομα ανεργίας, γιατί θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε εργασία. Επομένως υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου οι νομικές ε, ε, δεσμεύσεις είναι πολλές και όπου πραγματικά μπορεί να σημάνει μεγάλη αλλαγή ή οποιαδήποτε αλλαγή του νομικού πλαισίου. Το άλλο θέμα είναι η ποιότητα της θελοντικής προσφοράς. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες με δεσμευτική νομοθεσία ε, όπου ε, ασφαλίζονται έναντι τρίτων όλοι οι εθελοντές, οποιαδήποτε μορφή εθελοντικής εργασίας ε, και αν παρέχουν ε, και πρέπει να πω ότι χώρες όπως η Μακεδονία, ας πούμε, λέει ο μιλητής, ε, που δεν είναι βέβαια ακόμα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχει προχωρήσει ακόμα παραπέρα έτσι ώστε να προστατεύσει τους εθελοντές στη διάρκεια της παροχής εθελοντικής εργασίας. Το δεύτερο σκέλος της, του, του θέματος αυτού, του ζητήματος αυτού, είναι να διασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας εθελοντική εργασία. Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για τον χάρτη δικαιωμάτων ε, και υποχρεώσεων των εθελοντών. Τρίτη προτεραιότητα και μπορώ μόνο να συμφωνήσω με όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, θα πρέπει να διευκολυνθεί η εργασία ε, των εθελοντικών οργανώσεων. Νομίζω ότι ο καθένας από εμά που βρισκόμαστε εδώ έχουμε να διηγηθούμε μια οδυνηρή εμπειρία ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκολυνθεί η εργασία των εθελοντικών οργανώσεων, να μειωθεί η απίστευτη γραφειοκρατία και χαρτούρα από την οποία πρέπει να περάσουμε, ε, πράγματα που κάνουν εξαιρετικά περίπλοκο και χρονοβόρο ε, το έργο μας και με την διαδικασία γενικότερα όσον αφορά, ε, ε, και νομίζω ότι τώρα στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, του οικονομικού προγραμματισμού και πλαισίου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη προχωρήσει χώρες σε κάποιες νέες σε, σε, σε, κάποια, σε, σε κάποιες νέες διατάξεις, αλλά αυτές δεν είναι δεσμευτικές και δεν ισχύουν για όλες τις χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια κάθε νέας ευρωπαϊκής προτεραιότητας θα πρέπει να αναγνωριστεί και ένα σκέλος ε, εθελοντισμού. Ε, κάτι που αναφέρθηκε επίσης, ένα τέταρτο σημείο στο οποίο έχουν ήδη αναφερθεί προαλήσαντε, είναι η αναγνώριση και πιστοποίηση των, ε, ε, της γνώσης που αποκτούν και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι εθελοντές. θα πρέπει να, να υπάρξει ένας τρόπος έτσι ώστε να γίνουν ορατά ε, τα ε, ωφέλη που έχουν και οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι εθελοντές από τη μία πλευρά ε, και να γίνουν ορτά για τις επιχειρήσεις και εύκολα αναγνωρίσιμα αυτά τα στοιχεία, οι δεξιότητες κτλ. Ο κύριος Μερές ε, είπε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει η πρωτοβουλία ε, των, του Ευρωπαϊκού Έτους και πραγματικά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών αποκτά λίγο καλύτερη μορφή πλέον το έτος αυτό και πλέον πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για την υλοποίηση του έτους. Ερχόμαστε σε επαφή επομένως με όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Τίποτα ε, χωρίς εμάς πρέπει να είναι το σλόγγαν μας, ε, γιατί θα πρέπει να είμαστε παρόντες λοιπόν σε όλες τις διαργασίες ε, και όλες τις διαδικασίες. Ε, υπόθηκε και συμφωνώ ότι ο εθελοντισμός είναι οριζόντια διαδικασία. Ε, βεβαίως τα πράγματα μπερδεύονται λίγο γιατί δεν είναι σαφής ο καταμερισμός των ε, ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. Ε, πιστεύουμε ότι για να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε προβλήματα θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, διάλογος ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, στα εμπλεκόμενα μέρη, ανάμεσα στη κοινωνία των πολιτών μέσω των εκπροσώπων της και τους ε, ε, αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις ε, λήψης απόφασης. Δεν νομίζω ότι πολλές είναι οι κυβερνήσεις αυτές οι οποίες γνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εθελοντές και οι εθελοντικές οργανώσεις. Ε, μέχρι τώρα ε, ο διάλογος βασίζεται στον, στην ανοιχτή, στον ανοιχτό συντονισμό. Ενδεχομένως ε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τους οποίους μπορούμε να εφαρμόσουμε. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί ο διάλογος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η τοποθέτησή μας όσον αφορά τον εθελοντισμό. Επίσης, πιστεύουμε ότι ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και η οργάνωσή του ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια λευκή βίβλο με το ίδιο θέμα. Και τέλος, ε, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα, παρακαλώ πολύ ενεργήστε έτσι ώστε το τελικό κείμενο να γίνει δεκτό. Ξέρουμε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει ε, αλλάζουν οι διαδικασίες. Εμείς ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εξέλιξη αυτή γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό που το Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερες εξουσίες αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να ληφθούν τελικές αποφάσεις έτσι ώστε να διοργανωθεί σωστά το έτος αυτό. Τέλος, πιστεύω ότι δεν πρέπει απλά να μιλάμε για προβλήματα, διακυβεύματα, φραγμούς, δυσκολίες γιατί στο τέλος μιλάμε για 100 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, που είναι δεσμευμένοι, στρατευμένοι στον εθελοντισμό και που παράγουν έργο κάθε μέρα. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού θα είναι μια καλή ευκαιρία να χαιρετήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών και τη συμβολή τους στην κοινωνία μας επανερχόμενος σε προσωπικό επίπεδο, η ερώτηση στην οποία έπρεπε να απαντήσουν όλοι χθε Τι κάνατε την 9η Νοεμβρίου πριν από 20 χρόνια και δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να ε, απαντήσω. Ήμουνα προφανώς στο χωριό μου. Ε, δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι και θυμώνω που δεν θυμάμαι. Ε, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να θυμόμαστε τι κάναμε τη στιγμή που κάτι αξιοσημείωτο ε, συνέβαινε στην ε, ιστορία. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να ακολουθούνται από συγκεκριμένες και συνεκτικές δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πει, λέει η πρόεδρος, να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό η Σουηδική Προεδρία, το θέμα δηλαδή της ονομασίας του έτους. Ε, ε, αν πούμε τώρα ναι, απαντήσουμε ναι ή όχι, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την, το έτος αυτό. Μπορούμε να πούμε του χρόνου όχι, αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε το πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς αφού ο κύβος ερήφθη, ας κοιτάξουμε να ενεργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι παλαιοί κανόνες ε, δεν είναι τόσο ε, αυστηροί. Μας αφήνουν περισσότερη ευελιξία, γι' αυτό βιαστήκαμε να το ολοκληρώσουμε υπό Σουηδική Προεδρία. Ας αρχίσουμε τώρα από τον τελευταίο ομιλητή του προηγούμενου πάνελ και ας μιλήσει πρώτος. Ο κύριος Βελέμς. Ευχαριστώ πολύ. Όσα άκουσα βρήκα ότι είναι πολύ θετικά και μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όντως να συμμετέχουν περισσότεροι στην εθελοντική εργασία. Άκουσα για το γλωσσικό ζήτημα, ε, για το volunteering τι περιλαμβάνει, ότι περιλαμβάνει περισσότερα από αυτά που λέμε συνήθως. Λοιπόν, τρία πράγματα. Πρώτον, αναγνώριση είπαμε. Ε, επίσης, τα προσόντα, η κατάρτιση και τα θετικά για τους ίδιους τους εθελοντές. Μετά έχουμε την κοινωνία. Τι μπορεί ε, να πάρει η κοινωνία από αυτή την εργασία. Και έπειτα για τα στοιχεία όπως είναι το Youth Pass. Ναι, Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν θα πρέπει να τυποποιήσουμε υπερβολικά ώστε να καταλήξουμε σε μια νέα γραφειογραφία με σφραγίδες που πρέπει να μπαίνουν στα διάφορα χαρτιά. Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε ποιότητα. Και την ποιότητα μπορούμε να την πετύχουμε μέσω ε, της ε, ε, προσπάθειας που θα κάνουμε και μέσω των ευκαιριών που θα δώσουμε στους νέους και κυρίως εκείνους που δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο τους. ώστε να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Τώρα, τι προσόντα χρειάζονται. Αυτό δεν είναι προκαθαρισμένο. Πολλά και διάφορα προσόντα. Ποικιλομορφία υπάρχει και εδώ. Δεν υπάρχει μία κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να πάει η κοινωνία. Ένας άλλος τρόπος αναγνώρισης της εθελοντικής εργασίας είναι να περάσει λίγο και στο σχολικό κουρίκολουμ. Την προηγούμενη εβδομάδα που ζήτησα μισή μέρα άδεια για να έρθω εδώ, ε, και αυτό είναι συμβολικό βέβαια. Όταν πρόκειται για θελοντική εργασία. Κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει είναι η απλοποίηση του διοικητικού φόρτου και η εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνουμε στις εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στη Φλάνδρα, για παράδειγμα, οι οργανώσεις των νέων έχουν ε, το δικαίωμα να ε, για τρία χρόνια, να υποβάλουν διέτοιμα για τρία χρόνια και για τρία χρόνια να έχουν χρηματοδότηση και τα διοικητικά που ετοιμάζουν είναι κάτι θετικό και για αυτούς, γιατί τα ετοιμάζουν, φροντίζουν για την ποιότητα. Άκουσα πολλά ωραία πράγματα εδώ σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Williams. Ο κύριος Ρατσάνο. Allora, io condivido Κοιτάξτε, εγώ ε, συμμερίζομαι την ανάγκη ε, ταχύτητας. Πρέπει γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις. Και όπως λέμε και στην Ιταλία, καλύτερα να έχουμε το αυγό σήμερα παρά την κότα αύριο. Ε, και μην ξεχνάμε ότι σε ένα χρόνο, ο ένας χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια πραγματικά καλή δουλειά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα, ε, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε τον στόχο μας, θα, χάσουμε την εστίαση μάλλον. Σε σχέση με αυτά που είπε και η κυρία Κώστα πρώτη, αλλά που είπαν και άλλοι, ποιο, ποιος θα είναι ο ορισμός, ποια θα είναι η επικεφαλίδα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος δίπλα δηλαδή ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε τη λέξη βολονταριά, εθελοντισμός, ευρωπαϊκό ε, έτος εθελοντισμού. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στα γαλλικά, γιατί στα γαλλικά υπάρχουν δύο όροι και βεβαίως η, η σωστή περιγραφή είναι πάρα πολύ σημαντική παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία πρόταση που να, με τις να συμφωνούν όλοι. Ε, ο ορισμός λοιπόν κατά την άποψή μου μπορεί να είναι ε, μια παροχή υπηρεσιών ε, για την επίτευξη κοινού στόχου, κοινού κοινωνικού ωφέλους χωρίς ε, μετά από ελεύθερη απόφαση του ατόμου ε, και χωρίς οποιαδήποτε είδους αμοιβή. Βεβαίως δεν είναι το Ευαγγέλιο, είναι μια πρόταση που κάνω όσον αφορά τον ε, ορισμό. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι έχουν ληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες και μια βουλευτής η οποία έφυγε δυστυχώς ήταν από τους προτεργάτες Τη ε, ε, της ε, πρωτοβουλίας αυτής που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για την συνθήκη της Λισαβόνας και για την καθαρά νομική προσέγγιση. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τους τύπους, γιατί οι τύποι καμιά φορά είναι πολύ συσταλτικοί. Θα πρέπει λίγο να διευρύνουμε, νομίζω, τον ορισμό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μάλλον στο Συμβούλιο, όταν ε, το Συμβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει ε, και να υιοθετήσει την ε, πρόταση πιστεύουμε ότι θα πρέπει το κύριο μέλημά μας να είναι να επιτύχουμε το στόχο μας. Βεβαίως ο στόχος μας δεν είναι να πετύχουμε ένα καλό ευρωπαϊκό έτος ε, ε, εις βάρος των συνθήκων. Απλώς εγώ λέω ότι ε, μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλον, να αντλήσουμε πραγματικά ε, μεγάλο ε, κοινωνικό πλούτο, διαβάζοντας, δίνοντας μια νέα πνοή στις συνθήκες και βεβαίως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην καταδικάσουμε σε αποτυχία από την αρχή το ευρωπαϊκό έτος. Όσον αφορά τώρα τους διαγωνισμούς, ετέθη λοιπόν το ζήτημα αυτό που ξεπερνάει τον, ε, ε, την χρηματοδότηση των, ε, του περιεχομένου των διαγωνισμών. Ξέρετε, άλλο πράγμα οι προμήθειες, άλλο πράγμα οι διαγωνισμοί ακόμα και στις ε, προμήθειες και μάλλον ακόμα και στους διαγωνισμούς για τον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 για τον ομοιοδότη, ε, δεν ε, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να απλώς, όταν μιλάμε για το ειδικό αντικείμενο του εθελοντισμού, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε, οποιοδήποτε μπέρδεμα και παρεξήγηση. Πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν προς αποφυγή παρεξηγήσεων τι σημαίνει εθελοντισμός, ε, με ποιο τρόπο μπορούν, μπορεί η εθελοντική εργασία να συστρατευτεί κατά κάποιο τρόπο ή να συνυπολογιστεί ε, προς την εργασία των ε, επιχειρήσεων, να τα πούμε όσο γίνεται πιο συνολικά και όσο γίνεται πιο καθαρά. Ε, να μην ξεχωρίζουμε τα πράγματα, να μην τα κατακαιρματίζουμε έτσι ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο στόχος μας. Νομίζω Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ξεχάσουμε και να ξεπεράσουμε αυτές τις ιδέες οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί ότι δήθεν ε, οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει να συμβάλλουν κατά 20% στη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων ευρωπαϊκών. Δεν έχουν οι εθελοντές, δεν έχουν οι εθελοντικές οργανώσεις αυτά τα χρήματα. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί αυτό το 20%. Πάντως πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι πολύ ευτυχής με τη συζήτηση που έγινε σήμερα γιατί διαπιστώνω ότι Αντίθετα με, το, με την κατάσταση που προκρατούσε μερικά χρόνια πριν, στο Κοινοβούλιο και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το θέμα ε, του εθελοντισμού αρχίζει να εμβαθύνεται, αρχίζει να διευρύνεται και αρχίζει να γίνεται πιο κατανοητό. Έχει εμπλουτιστεί λοιπόν ε, η συζήτηση με νέα στοιχεία, ε, έχει γίνει πιο ευρεία και αυτό μας ικανοποιεί απολύτως. Τώρα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να καθορίσουμε ένα είδος μόνιμης στρογγυλής ε, τράπεζας όπου ε, θα, ε, κάνουμε μια, θα, θα προχωρήσουμε την συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα. Και πιστεύω ότι από αυτήν την άποψη όχι μονάχα ο οργανισμός τον οποίον εκπροσωπώ εγώ αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα είναι στην διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με μεγάλη ταπεινοφροσύνη να προσφέρουν την ε, συνεισφορά τους ε, στην συζήτηση αυτή. Επομένως υποβάλλουμε και στην Πρόεδρο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν την διαθεσιμότητά μας. Και τι να σας πω, Μέχρι τώρα ας πούμε ότι ξεφύγαμε με μία και ε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση αυτή, τη σκαπουλάραμε κατά κάποιο τρόπο μόνο με μία έκθεση. Ε, δεν γίνεται στο μέλλον όμως να συνεχίσει αυτό γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρατσόνη, ο κύριος Δικάπο. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για όσα μας είπαν. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σαμές γιατί μας έδωσε ε, πολλά σημεία επί των οποίων να σκεφτούμε. Εγώ ασχολούμαι, όπως σας είπα, πολύ με τον εθελοντισμό και την νεολαία ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ. Θα ήθελα να απομονώσω κάποιες ε, ερωτήσεις οι οποίες μου φάνηκαν ε, ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Πολύ μεταξύ ημών αναφέρθηκαν στην αξία του εθελοντισμού αλλά και στο περιεχόμενο του εθελοντισμού και νομίζω ε, Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ε, είπατε ότι αν διευρύνουμε την βάση συμμετοχής ε, τότε θα χαμηλώσει η ποιότητα. Ε, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Πιστεύω ότι η διεύρυνση της βάσης του εθελοντισμού μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Απλώς θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να παραμείνουμε ελεύθεροι, θα, ε, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις εμπειρίες, όλες τις εμπειρίες, ξεκινώντας από τις πάρα πολύ μικρές, τις μικρότερες, τις πιο μεγάλες και βεβαίως με λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά σίγουρα με κάποιους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν για όλους, που θα πρέπει να είναι ομοιογενείς. Η κυρία Κώστα αναρωτήθηκε για τον ρόλο ε, τον οποίον ε, ε, εγώ διαδραματίζω ως παίζω, ως διευθυντής αυτού του οργανισμού. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία ευθυγραμμίζεται με αυτά που συμβαίνουν και στις άλλες χώρες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει με μία δράση, στην οποία και ο κύριος Δάνεση προηγουμένως, ε, μία πολύ στοχευμένη ε, διαδικασία, ε, η οποία όμως δεν έχει αρκετή πρικοδότηση, αρκετή χρηματοδότηση και που βεβαίως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετή η κατεύθυνση λοιπόν προς την οποία ε, κινείται είναι ε, να ε, αναγνωριστεί η ποιότητα του παρέχοντος εθελοντική υπηρεσία και βεβαίως η αναγνώριση της ίδιας εθελοντικής υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς ζητούμε από τις οργανώσεις να υπάρχει ομοιογενές ενιαίο ποιοτικό επίπεδο ε, βάσει του προγράμματος νεολαία σε δράση και ε, κατά αυτήν την έννοια να ευθυγραμμιστούν σε αυτό δηλαδή το ποιοτικό επίπεδο να ευθυγραμμιστούν ε, και οι, οι, όλες οι οργανώσεις. Βεβαίως θα πρέπει να αφήσουμε τις οργανώσεις ελεύθερες να κινηθούν, βεβαίως θα πρέπει να αφήσουμε τους εθελοντέ ελεύθερους, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να διέπονται από κάποιους κοινούς κανόνες, γιατί οι κανόνες πάντα πρέπει να ε, υπάρχουν. Ε, και μετά βάσει και της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα να δοθεί δυνατότητα σε όσο γίνεται περισσότερους να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα. Ε, ρωτούσε η κυρία Κώστα με ποιο τρόπο μεταφράζονται αυτές οι αρχές σε δράσεις επιτόπου. Εγώ μπορώ να απαντήσω για την Ιταλία, αλλά ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς έχουμε την δέσμευση να προωθήσουμε την τις δράσεις μας, τις δράσεις αυτές και επίσης να υλοποιήσουμε δράσεις συγκεκριμένες οποτεδήποτε αυτό μας ζητάτε από το πρόγραμμα. Και οι οργανώσεις θα πρέπει να κάνουν τα προγράμματα πιο ορατά. Ε, επομένως, εμάς, μας, ε, ε, αυτό το ζητούμενο από μας είναι να κάνουμε πιο εμφανή, πιο ορατά τα αποτελέσματα, να ε, διαχέουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, τα αποτελέσματα. Γιατί τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά ε, ε, παράδειγμα σωστής υλοποίησης προγραμμάτων. Εμείς λέγαμε πριν ότι ο εθελοντισμός έχει μια πολύ έντονη τοπική διάσταση. Δεν υπάρχουν μονάχα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, εμείς δουλεύουμε σε μικρό τοπικό επίπεδο, σε μικρή κλίμακα, σε τοπικό επίπεδο. Δουλεύουμε ε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με μικρές τοπικές οργανώσεις. Και επίσης δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν ε, έχει καταβληθεί προσπάθεια από την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Ε, θα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν πραγματικά θέλει δηλαδή η Ευρώπη να ε, υλοποιήσει προγράμματα θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί και σε ε, νέους που δεν είναι στρατευμένοι και σε νέους που δεν εργάζονται ήδη μέσα στα πλαίσια οργανισμών, οργανώσεων ή σωματείων. Μέσω λοιπόν του προγράμματος νεολαία σε δράση ε, μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε νέους μέσα στα πλαίσια άτυπων ε, οργανώσεων ε, και επομένως οι νέοι αυτοί ξεκίνησαν ε, ξεκίνησαν κάποιες ε, οργανωμένες ε, δράσεις χωρίς να είναι μέλη σε κάποια οργάνωση και αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατά αυτή την έννοια βεβαίως χρειαζόμαστε και τη βοήθεια και την αρρωγή των τοπικών αρχόντων της τοπικής κοινωνίας, των τοπικά εκλεγμένων. Να σας πω ας πούμε ότι για πρώτη φορά φέτος οι δραστηριότητες για θέματα εθελοντισμού που θεωρητικώς κανονικά ε, χρηματοδοτούνται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είδαν Είδαμε ότι μετά από αίτημα της οργάνωσής μας ε, είχαμε επιπλέον κρατική ε, επιδότηση. Ας πούμε, εμείς είχαμε τέτοια επιπλέον χρηματοδότηση για δράσεις οι οποίες ανελήφθησαν στις ε, ε, περιοχές ε, οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή και επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, και άλλα πράγματα θα μπορούσα να σας πω, αλλά νομίζω ότι για να σεβαστώ τον χρόνο που είχα, θα πρέπει να ολοκληρώσω σιγά σιγά. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας και τα οικονομικά στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία. Βεβαίω αναφέρθηκε προηγουμένως ότι θα θέλαμε, θα επιθυμούσαμε από τους 3 στου δέκα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ε, να φτάσουμε στους 7 στους 10. Τα προγράμματα ε, τα οποία αφορούν την κινητικότητα των νέων είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί εκεί έχουμε την δυνατότητα να εμπλέξουμε τους νέους. Ε, γιατί ξέρετε, το, τα προγράμματα αυτά τελικά διαπιστώνουμε όταν κάνουμε τους τελικούς λογαριασμούς ότι ε, δεν έχουν απασχολήσει πάρα πολλούς νέους. Ε, και πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και το ανέφερα γιατί πραγματικά το πιστεύω, ε, ε, έφτασε να εμπλέξει, ε, μάλλον όχι, έφτασε να δώσει, να βοηθήσει έναν στους 100 από αυτούς που θα έπρεπε να αγγίξει. Το πρόγραμμα Έρασμους, το οποίο είναι το πιο αξιολογημένο και το πιο γνωστό τελικά καταφέρνει να δώσει, να ευεργετήσει 3% από τους ε, επιλέξιμους ε, δικαιούχους. Ε, και επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και το, το, το κύριο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η πληροφόρηση και η επικοινωνία. Γιατί Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Έτος είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ρίξουν οι προβολείς το φως τους ε, σε ανθρώπους που συνήθως εργάζονται στο σκοτάδι, που εργάζονται αθόρυβα και χωρίς κανείς να τους παίρνει ε, είδηση. Επομένως, πληροφόρηση και επικοινωνία. Και να μην ξεχνάμε ότι εάν οι δικαιούχοι της ε, αλλαγής, ε, δεν, οι δικαιούχοι ενός προγράμματος ε, δεν, καταλα... δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα αυτό, δεν το καταλαβαίνουν, άρα δεν έχουν κανένα ευεργέτημα, κανένα όφελος, ε, από το πρόγραμμα αυτό, τότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε αποτύχει και ότι η αποτυχία βαρύνει τους δικούς μας ώμους. Επομένως, θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία επιτόπου ε, ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με, την, με τον εθελοντισμό, τους νέους, τους λιγότερο νέους και από την άλλη μεριά αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτοί ακριβώς που παίρνουν τις αποφάσεις θα πρέπει να κατανοήσουν ότι μονάχα μέσα από το διάλογο, μέσα από την συνδιαλλαγή θα μπορέσουν και τη διαβούλευση θα μπορέσουν να Ολοκληρώνουμε αυτή την ακρόαση και έτσι θα ήθελα πρωτού δώσω τον λόγο στον κύριο Κορέα για να παρουσιάσει την έκθεσή του, πολύ σύντομα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι αυτό το θέμα της εθελοντικής υπηρεσίας είναι ένα θέμα το οποίο με μοναδικό τρόπο διεξάγεται και υλοποιείται εκεί όπου υπάρχει αυτό το όνομα και ο τίτλος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών. Πολύ σημαντική υπόθεση. Και για τον κύριο Ρατσάνο που είπε ότι τώρα θυμηθήκαμε και σκεφτήκαμε αυτό το θέμα να του πω ότι αυτή η υπηρεσία εθελοντών νέων ξεκίνησε με μια προφορική ερώτηση του συναδέλφου μου Αλεξάνδερ Λάνε από τον Νότιο Τυρόλο. Και εμείς με μια προφορική λοιπόν ερώτηση προωθήσαμε αυτό το θέμα κύριε. Και κατά τα άλλα σε σχέση με την άτυχη επίτροπο Κρεσόν προήχθη τότε επ' αυτής της θητείας. Αν παραμένει κάτι, παραμένει η εθελοντική υπηρεσία νέων από τότε. Και ήταν μια ιδέα της Ευρωβουλής, βλέπετε, του Αλεξάνδρου Ελάγα και της Ντόχρης Πακ από δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αλλά με μεγάλες προσπάθειες υπέρ των νέων. Θέλω να το πω αυτό, καμιά φορά πρέπει να αυτό επενείται κανείς, γιατί ε, πρέπει να πενέσει στο σπίτι σου, μην πέσει και σε πλακώσει. Λοιπόν, πάνε χρόνια τώρα γι αυτό, από αυτό και το καταφέραμε. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η υπηρεσία εθελοντών νέων όχι μόνο κατά το έτος της ε, Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει να προσεχθεί, αλλά και σε πολλούς τομείς πολιτικών που στο εγγύς μέλλον θα δούμε και θα εξετάσουμε. Στο πρόγραμμα για την νεολαία θα διαδραματίσει ένα ρόλο, αλλά επίσης και στην ε, εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων θα διαδραματίσει και πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Και για το θέμα της νεολαία των νέων επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στον τομέα της ολοκλήρωσης, ενοποίησης ολοκλήρωσης. Δεν χρειαζόμαστε μόνο νέους που όπως ο συνάδελφος ε, Ρατσάνο προανέφερε ο Επαϊόν, νέο δεν θυμάμαι ποιο το είπε, για νέους ε, που δεν μπορούν να μεταβάλουν προσπάθειες επειδή λέει να ετούνται σε άσυλο, αλλά χρειαζόμαστε εκείνους τους νέους που είναι εδώ, και αν δεν μπορούν να εργαστούν και δεν έχουν εργασία σε τακτική σχέση απασχόλησης, τότε εθελοντικά θα μπορούν να απασχοληθούν και να καταβάλουν προσπάθειες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής της κοινωνίας. Θα είναι και για αμφότερες τις πλευρές ε, εποφελές. Χρειαζόμαστε και νέους ενήλικες που θα βοηθήσουν αυτούς τους νέους και θα συνεισφέρουν. Είναι ένα θέμα αμοιβαιότητας και πρέπει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων, στα επόμενα προγράμματα να λάβουμε αυτό υπόψη. Ένα πράγμα θέλω να υπενθυμίσω. Ένας Έλληνας συνάδελφος είναι εδώ. Υπενθυμίζω αυτές τις τρομερές πυρκαγιές, δασοπυρκαγιές στην Ελλάδα. Θέλω να υπενθυμίσω και να πω, αν στην Ελλάδα υπήρχαν πολλές πυροσβεστικές υπηρεσίες και εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, εθελοντών πυροσβεστών, όπως σε άλλες χώρες, πολύ καλύτερα θα καταπολεμούσαμε τη φωτιά τότε. Δεν θέλω κανένα να κατηγορήσω. Είναι μια, μια παράδοση, έχουμε μακρά χρονική παράδοση στη Γερμανία εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών. Και είναι σημαντικό αυτό. Και ακριβώ οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ελλάδα θα χρειαζόντουσαν έντονα και θα ήταν πολύ χρήσιμοι. Αλλά και αλλού, εκεί όπου υπάρχουν πυρκαγιές και δεν υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες. Υπάρχουν πολλοί τομεί λοιπόν σίγουρα όπου ο εθελοντικό τομέα, ο ρόλο τη εθελοντική εργασία έχει μεγάλη σημασία. Ένα συνάδελφο αναφέρθηκε στα αθλήματα. Έχουμε τα αθλήματα τώρα στη συνθήκη. Δώσαμε αγώνα γι' αυτό. Τώρα το έχουμε. Κατοχυρώνται στι συνθήκε. Και έχουμε τον εθελοντικό χαρακτήρα τη συμμετοχή. Χρειάζεται ο εθελοντικό χαρακτήρα, η βούληση αυτή και η αναγνώριση του ρόλου των εθελοντών. Πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Χρειαζόμαστε μια πιστοποίηση, μια αναγνώριση όπως και αν διαμορφωθούν τα πράγματα. Μπορεί να είναι διαφορετικά σε εθνικά πλαίσια αυτή η πιστοποίηση, η αναγνώριση, αλλά πρέπει να υπάρχει και να αντανακλάται στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ευρωπαϊκά, ώστε οι νέοι να μην μπορούν μόνο να πούν ότι «Α, έχω αυτό το πιστοποιητικό αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, αλλά έχω ένα πιστοποιητικό σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, κοινωνική υπηρεσία που προσέφερα. Αυτό είναι μια σκέψη και σε σχέση με την από τότε που ιδρύθηκε η Ευρώπη ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να γεμίσουμε με περιεχόμενο τέτοιες προτάσεις. Έχουμε πάμπολες ιδέες που ελπίζουμε ότι αυτές οι ιδέες πριν από το έτος των εθελοντών θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και ίσως και κατά τη διάρκεια του έτους εθελοντών να μπορέσουν να προαχθούν, να αναζωογονηθούν και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ όλους εξ ονόματος των συναδέλφων τους επαίοντε που ήταν εδώ παρόντε, που ήταν τόσο ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσει τους και οι εισηγήσει τους και έδωσαν αρκετές απαντήσεις και σε μη διατυπωμένε <laughs> ερωτήσεις αλλά και σε θέματα που είχαν τεθεί από εμάς. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε, ο κύριος Κορέα θα λάβει τον λόγο για να μπορέσει να μα παρουσιάσει τα, τη του. Παρακαλώ κύριε Κορέα, έχετε τον λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους τέσσερις εμπειρογνώμονες ε, εισηγητές που ε, μας οδήγησαν σε μια ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρέπει να πω ότι αυτή η συζήτηση που έλαβε χώρα ε, κατέστησε σαφή δύο πράγματα. Πρώτον, την μεγάλη ανάγκη όχι μόνο να μιλήσουμε, αλλά να ε, αντιμετωπίσουμε με τον πλέον ευρωπαϊκό τρόπο το ε, θέμα αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, η μεγάλη διαφοροποίηση εμπειριών στα, στις διάφορες χώρες, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή βλέπουμε ε, ότι στη Γαλλία ας πούμε η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Εκεί υπάρχει και η διαφορά που δεν υπάρχει σε άλλες χώρες ανάμεσα σε μπενεβολά και βολονταριά. Ε, φτάνουμε ε, στην ε, Ιταλία η οποία ξεχωρίζει τον εθελοντισμό από, τα, από τους κοινοφελείς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ε, βλέπουμε λοιπόν μια, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Εν πάση περιπτώσει κατανοούμε, διαπιστώνουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να εναρμονίσουμε αυτές τις διαδικασίες γιατί ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο κίνημα ε, εθελοντισμού ε, και είναι κρίμα η Ευρώπη μας να μην ε, ασχοληθεί ακόμα περισσότερο με τον εθελοντισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση κάποιων, στη διάθεση του, του, κοινού καλού, στη διάθεση του κοινού ωφέλους. Ε, και νομίζω ότι κατά αυτήν την ε, έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον εθελοντισμό και να εναρμονίσουμε ε, τα, του εθελοντισμού. Ε, επίσης, σήμερα ασχοληθήκαμε και με το πολύ συγκεκριμένο πράγμα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό έτος ακριβώς δημιουργείται, ε, θεσμοθετείται έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη ε, για το θέμα αυτό ε, και αφετέρου ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο καλύτερο να λειτουργήσει ο εθελοντισμός ε, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ακόμα και ε, νομοθετικές διορθώσεις, έτσι ώστε οι εθελοντές, έτσι ώστε οι εθελοντικές οργανώσεις, όποια μορφή και αν ε, υφίστανται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να, να αποκτήσουν μια πιο ενιαία ας πούμε, δράση και αντιμετώπιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο, όπως το έκανα και σήμερα το πρωί άλλωστε, αλλά και το, την ε, προεδρία, τη Σουηδική Προεδρία, η οποία δια του εκπροσώπου της ε, κάθισε στο ίδιο τραπέζι μαζί μας ε, και μπορέσαμε να συζητήσουμε από κοινού κάποια πράγματα, να συμμεριστούμε κάποιες απόψεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια καλύτερα πράγματα. Είναι αλήθεια και το είπε κάποιος ομιλητή προηγουμένως ότι κάλιο, 10 και στο χέρι, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και να τα περιμένουμε για κάποια χρόνια. Επομένως, ας ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι δεδομένα ε, για τώρα και αργότερα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα εγώ να μιλήσω μονάχα για ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μου δεν ε, συζητήθηκε αρκετά, δηλαδή το όνομα αυτού, αυτού του έτους. Μιλάμε για Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, αλλά οι υπηρεσίες μας λένε ότι στην ουσία το να μιλήσουμε για εθελοντισμό ε, με τόσο άμεσο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, γιατί ο εθελοντισμός τυπικά τουλάχιστον και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα βοηθήσει. Είναι ένα πολύ γενικό και ομό κατά κάποιο τρόπο ε, όνομα ε, το οποίο δεν είναι προτιμητέο. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ε, εθνι... Ε, ένα ευρωπαϊκό έτος για τις δράσεις οι οποίες είναι κοινωνικά οφελείς, εποφελείς και οι οποίες οδηγούν σε μια κοινωνική ευαισθητοποίηση. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένας περίεργο τίτλο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε λίγο πώ μπορούμε να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Ε, κατά την άποψή μου αυτός ο τίτλος που ανέφερα προηγουμένως είναι λίγο ε, ε, εκφοβιστικός και επομένως νομίζω ότι καλό θα ήταν αν μπορέσουμε να κρατηθούμε σε αυτό το, το, αρχικό έτος εθελοντισμού ή εθελοντικής προσφοράς ή τέλος πάντων κάπως να το πούμε με ένα πιο απλό τρόπο. Στις πρώτες τροπολογίες μου θα δείτε, διαβάζοντας το κείμενο, θα δείτε κάποιες ε, πρώτες, κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία θεωρώ ε, ε, σημαντικά και με τα οποία θα πρέπει, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι ε, και λαμβάνοντα υπόψη τι συζητήσει που έλαβαν χώρα μέχρι τώρα και λαμβάνοντα υπόψη του τύπου, ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε τι σημαίνει εθελοντισμό, τι εννοούμε με τον εθελοντισμό. Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα ανοιχτό θέμα, είναι μια ανοιχτή συζήτηση, η οποία βεβαίω οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κοινό υπόβαθρο. Ο καθένα αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό όταν μιλάει για εθελοντισμό και επομένω θα πρέπει να, να, να ε, ε αμβλύνομαι τις ε, παρεξηγήσεις ε, ή τις ε, διαφορές. Βεβαίως είναι γεγονός ότι η πρόθεση, ο σκοπός, ο στόχος του εθελοντισμού θα πρέπει να είναι η κοινή ωφέλεια, θα πρέπει να είναι ένα κοινωνικό έργο, θα πρέπει να είναι ένα πολιτιστικό έργο και επίσης θα πρέπει να αποτελεί ένα επιπλέον ε, στοιχείο για την ε, κοινωνία των πολιτών. Ε, θα πρέπει να είναι σαφές επίσης ότι η εθελοντική εργασία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να πάρει τη θέση αμοιβόμενης εργασίας, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει αμοιβόμενη εργασία, επαγγελματική εργασία. Και εδώ βεβαίως μπορεί να υπάρξει χώρος για μια περαιτέρω ε, συζήτηση, έστω και αν εγώ έχω ήδη υποβάλει τις ε, τροπολογίες μας. Έχουμε 48 ώρες ακόμα, αν έχετε 48 ώρε αν θέλει κάποιο να υποβάλει κάποια ε, ε, τροπολογία, αλλά ακόμα και μεταξύ μα μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι την επόμενη ε, εβδομάδα βέβαια θα έχουμε μια συνάντηση στο Στρασβούργο, αλλά ε, εγώ θέλησα να συναντηθούν ε, οι σκιώδεις ηγητές και η υπεύθυνοι γνωμοδότησης άλλων επιτροπών, έτσι ώστε να κάνουμε ομαδική εργασία. Νομίζω ότι εμείς νομίζω ότι υποχρεώσαμε όλους τους εμπλεκόμενους ε, να εργαστούν ε, με εξαιρετικά ε, δύσκολους και γρήγορους ρυθμούς, γιατί δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπορούμε να μαζευόμαστε και να δουλεύουμε όλοι μαζί. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλησα να υπογραμμίσω είναι ε, αυτό των δραστηριοτήτων. Διακινδυνεύουμε μερικές φορές, ε, ε, μάλλον, συγγνώμη, διατρέχουμε τον κίνδυνο μερικές φορές, τα ευρωπαϊκά έτη να είναι ευκαιρία για μεγάλες διασκέψεις, για πολλά και μεγάλα και παχιά λόγια. Ε, και ξεχνάμε λίγο τις, την, την πράξη και ξεχνάμε λίγο ε, τα έργα. Εγώ γι' αυτό το λόγο ακριβώς θέλησα να ε, ε, καταδείξω ότι η κατάσταση για το ευρωπαϊκό του εθελοντισμού θα πρέπει να είναι διαφορετική. Γνωρίζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια μελέτη για τον εθελοντισμό ήδη ε, στα τέλη τρέχοντος έτους ε, και επομένως μπορεί να υπάρξει επικάλυψη των διεργασιών. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θεωρήσαμε ότι στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης ε, αλλά και αξιοποίησης ε, των εθελοντικών οργανώσεων ε, και των ιδίων των ε, εθελοντών. Ε, θα πρέπει να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να αντιπαραθέσουμε επιτόπου τις δραστηριότητες διαφόρων οργανώσεων και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο και λόγω της φύσης του θέματος να αποφύγουμε τις μεγάλες διασκέψεις, τα μεγάλα συνέδρια ναι, φυσικά να έχουμε συναντήσεις ε, όπου ε, θα καταδειχθούν οι καλές ε, πρακτικές. Βεβαίως να, υπάρχουν, να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί νέα δυναμική σε αυτές της ινσίτου του δραστηριότητες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτό το ευρωπαϊκό έτος θα πρέπει να αφιερωθεί ε, σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, είτε πρόκειται για ε, πάροχους εθελοντικής εργασίας, είτε πρόκειται για αποδέκτες ε, εθελοντικής εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος έχουμε και την καυτή πατάτα του προϋπολογισμού. 6 εκατομμύρια ευρώ συν 2 ε, ε, εκατομμύρια ε, για το έτος 2010 ως έτος προετοιμασίας. Αυτά είναι τα χρήματα, αυτή είναι η χρηματοδότηση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά προηγούμενα έτη. Να σας πω, για παράδειγμα, ότι το έτος 2010, που είναι το έτος της μάχης ε, κατά της ε, Ένδειας, αν θυμάμαι καλά, έχει μια προκοδότηση τάξης των 17 εκατομμυρίων. Επομένως, ε, θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούμε με τόσο στριμωγμένα οικονομικά να ε, κάνουμε κάποιες ε, ε, δραστηριότητες και να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες βεβαίως θα είναι αποκεντρωμένες αλλά θα έχουμε και ένα τμήμα κεντρικό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα για πολλαπλές δραστηριότητες τα χρήματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι το 80% της 100 ε, των προγραμμάτων που αποτελεί παραδοσιακά συγχρηματοδότηση, ενδεχομένως και παραδόξως μάλιστα θα έλεγα, μπορεί να ε, δυναμητιστεί γιατί, ε, και για γιατί έχει γίνει ήδη μία πρόταση το, το ποσοστό αυτό να είναι της τάξης του 65%. θα δούμε, θα δούμε μέχρι το τέλος πώς ε, θα διαμορφωθεί ο προπολογισμό ε, και τι κονδύλια θα έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντως να φτάσουμε τουλάχιστον στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ήταν το ευκταίο, γιατί είναι πάρα πολλές δραστηριότητες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε το βασικό, τον βασικό προϋπολογισμό Ε, και νομίζω ότι είναι σαφές και έχει καταδειχθεί ότι το Κοινοβούλιο ζητάει υψηλόφωνα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, να ε, δοθούν περισσότερα χρήματα σε, το, σε αυτό το, το πρόγραμμα έτσι ώστε σαν ευρωπαϊκό έτος να έχει ε, όλες τις προϋποθέσεις να επιτύχει έχοντας έναν καλύτερο ε, προϋπολογισμό. Αυτά, αυτά εντάχει έτσι κι αλλιώς έχουμε το γραπτό, έχετε το γραπτό κείμενο, μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο γραπτό ε, κείμενο το οποίο έχετε στην διάθεσή σας. Ε, στο γραπτό κείμενο αναφέρομαι στη σημασία του εθελοντισμού, στον ρόλο που πρέπει να παίζει στην κοινωνία και στην κοινωνία των πολιτών. Γίνεται αναφορά στην επικουρικότητα, γίνεται αναφορά σε επιμέρους ε, σημαντικά θέματα. Ε, τώρα δεν θα σας διαβάσω όλο το έγγραφο, γιατί νομίζω ότι ακούσαμε ήδη πολλά θέματα, πολλά πολλά σκέλη αυτού του προβλήματος και επομένως δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκούρια. Έχω τώρα τον κύριο Φλίγεστάιν στον κατάλογό μου. Δεν ξέρω και αν κάποιοι άλλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα αρχίσουμε τον κύριο Φλιγεστάιν. Θα είμαι σύντομο και πιο πριν είχα πει κάτι. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εσάς κύριε Κορέα. Θερμά να σας ευχαριστήσω για την περιεκτική διεξοδική έκθεση που μας παρουσιάσατε. Οι προτάσεις στοχεύουν στη σωστή κατεύθυνση και σε μεγάλο βαθμό τις υποστηρίζουμε τις προτάσεις αυτές εμείς. Το Ευρωπαϊκό Έτος όχι μόνο πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να ε, ε κάνουμε δεκα, βγάζουμε δεκάρικους λόγους, Ανέφερα ότι είχα εργαστεί σε αυτόν τον τομέα και δεν έχω καμιά ανάγκη σε αυτή τη ζωή ε, να ακούω δεκάρικους λόγους. Περιτεύουν απόλυτα αυτοί. Κάτι αηφόρο πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό υποστηρίζω την πρότασή σας να δημιουργηθεί ένα μητρό, μια τράπεζα δεδομένων για την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, του εθελοντισμού και η αύξηση του προϋπολογισμού του κονδυλίου σε 10 εκατομμύρια. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω, όπου θα ήθελα μια συμπλήρωση να επιτευχθεί επιθυμώ να υπάρξει συμπλήρωση. Και σε ένα σημείο παρακαλώ να ξανασκεφτείτε τη θέση σας, την τοποθέτησή σας. Αφενός το είχα πει και πιο πριν. Μου φαίνεται ενδεδειγμένο εργα... εργαζόμενοι και συνδικάτα και ε, να μπορέσουν και οι εργοδότες να συμπεριληφθούν σε αυτή την ε, ε, εκδήλωση, ώστε το θέμα του εθελοντισμού και της έναντι αμοιβή εργασίας να αποτελέσει αντικείμενο ευαισθητοποίηση, να συνειδητοποιήσουμε τα πράγματα και να τα συζητήσουμε. Δεύτερον, θεωρώ την πρότασή σα για την συγχρηματοδότηση από 80% να μειωθεί η συγχρηματοδότηση σε 75%. Αυτή την πρότασή σας δεν τη θεωρώ πολύ καλή. Κατανοώ γιατί το κάνατε, για να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες το κάνατε. Αλλά από την εργασία μου, ε, ε, το έργο μου στην ε, Λιθουανία και τη Λετωνία και από άλλα μέρη, ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να δομήσουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, τον εθελοντισμό δηλαδή, να βρουν κονδύλια. Και θα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αν μέχρι 80% αν είναι αναγκαίο το 80% εκεί όπου είναι αναγκαίο το 80% να καλύπτεται έτσι και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο ε, ίσως ε, να καλύπτονται έτσι οι ανάγκες τους όχι 75 αλλά 80% λοιπόν. Και να διασφαλίσουμε επίσης, και είναι παράκλησή μου σε σχέση με την Ευρωβουλή και την κοινοβουλευτική μας ομάδα, οι δραστηριότητες αυτού του έτους εθελοντισμού να τις συνοδέψουμε και να τις παρακολουθήσουμε από κοντά, εκ του σύνεγγυς. Και όχι μόνο να έχουμε μια ωραία έκθεση, αλλά να συνδιαμορφώσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάω εκ μέρου της Μαρία Σάκη, τη συναδέλφη, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να μεταφέρω κάποια δικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστεί πολύ τον κύριο Σκούρη για τη δουλειά του και φυσικά και περιμένει να έχουν ανταλλαγή απόψε και μεταξύ τους. Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα λέει, που μπορεί να υποστηρίξει στην έκθεση για την κοινότητα που είναι μια κοινότητα αξιών, για το ρόλο των Ευρωπαίων πολιτών στον κόσμο, επίσης για τη συμμετοχή τη, του κόσμου στις δραστηριότητες, στις εθελοντικές που βοηθούν την κοινωνική συνοχή κλπ. Συμφωνεί επίση με τον κύριο Σκούρια για το ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια. Συνολικό προπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το ελάχιστο προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το ευρωπαϊκό έτο. Πιστεύει ότι τα ποσά τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί ε, για τα διάφορα ευρωπαϊκά έτη είναι τέτοια που και εδώ μα αναγκάζουν να ζητάμε 12 εκατομμύρια καλύτερα. Το θέμα αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά. Επίση, να χρησιμοποιηθούν τα μέσα επίσης για τα αλλαγή βέλτιστων ε, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι εθελοντές για να μπορέσουν να μοιραστούν την εμπειρία τους και ακόμα και πέρα από τα σύνορα τη Ευρώπη. Τα νέα μέσα ε, χρήσιμο μπορούν να προσφέρουν μάλλον πολύ περισσότερες δυνατότητε για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρών. Έχει βέβαια και διάφορε ερωτήσεις που θα σας θέσω εγώ εκ μέρου τη. Πρώτον, ο εισηγητής έχει να προτείνει κάτι για αυτό το πόρταλ, την πύλη τη, στο διαδίκτυο, ώστε, να νιώσουν οι θελοντές περισσότερο ε, δικιά τους αυτή τη ε, δουλειά του θελοντισμού και το έτος θελοντισμού. Δεν πρέπει να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης ανά τον κόσμο. Πολλοί Ευρωπαίοι είναι θελοντές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό συζητήθηκε βέβαια και πριν και είπαμε ότι είναι ένα από τα προβλήματα για ορισμένες χώρες τουλάχιστον προκειμένου να υπάρξουν εθελοντές. Μια άλλη ερώτησή της λέει ότι η συγγητής με σαφήνεια λέει ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα επιχειρησιακό πλαίσιο και όχι ένα νομικό πλαίσιο. Πιστεύει η συγγητή ότι υπάρχουν περιθώρια να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τις βέλτιστες πρακτικές όταν πρόκειται για θέματα που αναφέρθηκαν σήμερα όπω είναι οι συντάξει κλπ. Τέλος. Ρωτάει για την συγχρηματοδότηση. Υπογραμμίζει ο εισηγητής ότι θέλει περισσότερη χρηματοδότηση. Είναι καλή αυτή η φιλοδοξία βέβαια, αλλά να ρωτιέται αν λαβαίνει υπόψη εισηγητή στον κίνδυνο. Αν δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, εθελοντικέ οργανώσει που δουλεύουν με πολύ χαμηλό προπολογισμό ή χωρί καθόλου θα μπορούν να συμμετέχουν. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι να αποκλειστούν αυτοί που δεν μπορούν να συνεισφέρουν με το ποσοστό που πρέπει στον προπολογισμό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις της συναδέρφου. Εγώ θα έλεγα 75% αλλά πρέπει να ξέρετε ότι άλλοι σκιώδεις στην Κοινωνική Επιτροπή δεν το δέχτηκαν. Ίσως όμως θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα 10 ή 12 εκατομμύρια που ζητάμε, οπότε τότε το 80% της χρηματοδότησης θα μας επιτρέψει μια καλή κατανομή των πόρων. Η ανησυχία μας είναι ότι σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά σε χρηματοδότηση, αν είναι παραπάνω, θα τους δυσκολέψουν τη ζωή. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί, μπορεί, γιατί δεν ήμουν εδώ όλο το απόγευμα. Ρωτάω, το χρονοδιάγραμμα έχει οριστικοποιηθεί Είμαστε σίγουροι ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου που θα τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ξέρω την απάντηση. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Το αναφέραμε σήμερα το απόγευμα εδώ τη δυνατότητα της υπηρεσίας ε, της εθελοντικής των seniors. Αν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιδέα. Και τώρα έρχομαι στο τελικό μου σχόλιο, λέει η ομιλήτρια. Οι προσδοκίες για το ευρωπαϊκό έτος είναι τεράστιες. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε μερικά πράγματα το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, να φροντίσουμε να τα κάνουμε μετά, δηλαδή να επηρεάσουμε την πολιτική να αλλάξει κατεύθυνση σε αυτό το θέμα. Και οι εθελοντές από ολόκληρη την Ευρώπη έτσι να δουν ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις από την πλευρά μας, ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από αυτό το ευρωπαϊκό έτος, πέρα από την αναγνώριση των εθελοντών, του έργου τους κλπ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κώστα είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή γιατί πραγματικά προσπαθεί να λάβει υπόψη όλη αυτή τη διαδικασία παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και πολλές δυσκολίες. Πάντως με πολύ ενδιαφέρον τον άκουσα. Εγώ θέλω δύο πράγματα να πω. Πρώτον, για το, την ορολογία. Θα ήθελα να συμπεριλάβουμε όλες τις μορφές εθελοντισμού. Κατά τα άλλα έχω ακούσει βέβαια πάρα πολύ προσεκτικά. Πρέπει να δούμε νομικά τι πρέπει να αποφασίσουμε. Άκουσα και τον κύριο Ρατσάνο. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει και μια επεξήγηση. Βασικό πάντως είναι να είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό για την ονομασία του έτους. Δεύτερο, ένα πιο πολιτικό ζήτημα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να στριμωχτούμε νομικά και να περιορίσουμε ε, τους ε, εθελοντές. Αντίθετα, το ακούσαμε και από τους ομιλητές για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν εδώ οι προσκεκλημένοι μας. Το έτος αυτό δεν μπορεί να είναι ένα έτος που έχει φιλοδοξίες δραστηριοτήτων αλλά ελάχιστα κονδύλια. Όχι. Γιατί πρέπει να υπάρξει και η διάδοση των ε, βέλτιστων πρακτικών, αλλά πρέπει να έχει και μια πιο πολιτική χρειά για να έχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε στη λευκή βίβλο της Επιτροπής. Θα ήταν ενδιαφέρον στην έκθεση του Κοινοβουλίου να ζητάμε από την Επιτροπή πέρα από την πρώτη έρευνα αυτή που σίγουρα είναι πολύ σημαντική, να... Καλό είναι να έχουμε ομοιογενή στοιχεία βέβαια, δεν λέω, αλλά είναι σημαντικό να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω. Το έτος αυτό να θέσει τις βάσεις για μια διαδικασία μια κατεύθυνση. Δεν ξέρω πώς θα διατυπωθεί και ποιο θα είναι σωστό, αλλά να λέμε ότι ξεκινήσαμε με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για τον Αθελοντισμό, μετά να δούμε ποια είναι η νομοθεσία που έχει στα διάφορα κράτη-μέλη και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε, αν όχι σε μια ομοιομορφία, αν μη τι άλλο σε ένα στάνταρτο ορισμό, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε το καθεστώς εθελοντισμού που υπάρχει στις διάφορες χώρες. Κάτι άλλο για το οικονομικό. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια για περισσότερα κονδύλια. Όπως σωστά λέει και ο κύριος Σκούρια. Γιατί τα χρήματα που έχουμε τώρα δεν φτάνουν. Το 25% μπορεί να είναι πολύ για ορισμένους. Που ίσως πρέπει να πούμε μέχρι αυτό το ποσοστό και όχι να βάλουμε νούμερο. την ε, προτεραιότητα πάντως πρέπει να τη δώσουμε και στις μικρές οργανώσεις που έχουν μικρά project. Να μην τα αποκλείσουμε. Το άλλο ζήτημα, το άλλο ερώτημα είναι το εξής. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να να βάλουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος όλες τις επιθυμίες και όλα τα στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να περιλαμβάνει ο εθελοντισμός όμως ε, θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια mainstreaming το, Ευρωπαϊκό, το, ταμείο, το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο μπορεί, ε, και το ξέρω γιατί εγώ ε, υπήρξα διαχειρίστρια στην δικιά μου περιοχή, μπορεί να οργανώσει δημόσιες προμήθειες ή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, διευκολύνει τα πράγματα για τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις. Και επίσης μπορεί μέσω των κονδυλίων και του τρόπου διαχείρισής τους να υπάρξει αναγνώριση της προσπάθειας των ε, εθελοντών. Επομένως, νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε μία ευρύτερη, ας πούμε, έποψη. Και πρέπει να δούμε τι ε, γίνεται με τις ε, είδαμε τι έγινε και με τις γυναίκες. Ξεκινήσαμε από την ε, ίδια αμοιβόμενη εργασία και φτάσαμε στο mainstreaming σε όλα τα προγράμματα και σε όλα τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κίλεν ε, μετά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πρέπει και να ολοκληρώσουμε. Γιατί θα έχουμε και την Επιτροπή και τον κύριο Σκούρια ξανά. Και πρέπει να τελειώσουμε. Παρακαλώ κύριε Κέλλη. Δεν θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στους ομιλητές. Και χαίρομαι που ήμασταν τόσο πολύ. Πρέπει να το πούμε. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο 14 Ιουλίου, κατάλαβα ότι πολλοί ομιλητές θέλουν να περιορίσουν τη γραφειοκρατία στο Κοινοβούλιο. Και αυτά που ακούσαμε σήμερα ελπίζω να ληφθούν υπόψη και να υπάρξει δράση για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας κυρίως. Κάτι άλλο που δεν μπορούμε να αγνοούμε είναι το θέμα της ηθικής. Πολλές χώρες, όχι μόνο η δικιά μου, έχει δει καταχρήσεις να γίνονται. Ορισμένοι θελοντές καταχρώνται τις θέσεις τους. Αν υπάρχει και γραφειοκρατία, είναι δύσκολο να εντοπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα για την αύξηση του προπολογισμού. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος, πρέπει να φροντίσουμε να είναι και καλό. Άρα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Και το θέμα των εθελοντών δεν σταματάει βέβαια το 2011. Καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται και μετά. Οι εθελοντές είναι εθελοντές Διαβίωση συνήθω, όχι μόνο ένα χρόνο. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ένα καλό έτος εθελοντισμού. Οπότε τον τίτλο πρέπει να το προσέξουμε πολύ, να είναι απλό. Για τόσο πιο περίπλοκο θα είναι, τόσο πιο περίπλοκο θα είναι να βρούμε θελοντές. Όσο πιο απλό είναι ο τίτλο του έτου αυτού, τόσο πιο απλό και κατανοητό θα είναι και το μήνυμά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τέιλιν, επόμενη. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους εισηγητές που πήραν το λόγο σε εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων. Για τον τίτλο τώρα. Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο τίτλος. Και γιατί. Γιατί αυτό το έτος θα μας επιτρέψει ακριβώς να διευκρινίσουμε τις δραστηριότητες εθελοντισμού στις διάφορες χώρες, ανάλογα με την νομοθεσία που ισχύει στην κάθε χώρα. Δεύτερο, θέλω να επιμείνω για το ότι η εθελοντική εργασία μέσα σε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν πρέπει να αντικαθιστά μία αμοιβόμενη θέση εργασίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και ακόμα και οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τον εθελοντισμό για να αντικαθιστούν με ελάχιστο δυνατό κόστος έναν μισθωτό. Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, λοιπόν, το είπατε και εσείς κύριε Σίγητα, είναι για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη η ενίσχυση της ειρήνης, της συνεργασίας, ε, των σχέσεων Βορρά-Νότου. Ουσιαστικά είναι για να ε, απαλληφθούν οι διακρίσεις σε βάρος ορισμένων. Τέλος, θέλω να ενθαρρύνω τον εισηγητή και την έκθεσή του για να πω ότι οι εθελοντές πρέπει να υποφελούνται από μια προστασία και όσον αφορά την υγεία τους αλλά και όσον αφορά την ασφαλειά τους. Πόσοι και πόσοι δεν πάνε σε εργοτάξια ε, αμοιάντου. Πρέπει να προστατεύονται. Και όλα αυτά πρέπει να τα πούμε και να τα καταδείξουμε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου τώρα. Ελπίζω να πρόφερε καλά το όνομά σας, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Σκούρια και όλους τους εκπροσώπους από τις οργανώσεις που είναι σήμερα μαζί μας. Πραγματικά η εισήγηση του κύριου Σκούρια είναι εξαιρετική και συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των κονδυλίων είναι απαραίτητη. Ε, δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Θα το κάνω όμω επειδή αναφέρθηκε το παράδειγμα τη Ελλάδα και έχω και ένα ακόμη παράδειγμα εγώ να καταθέσω ελληνικό. Σε ό,τι αφορά την κατάσβεση των πυρκαγιών που είπε προηγουμένω η κυρία Πακ, το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από τον καθένα ότι η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς είναι μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη υπόθεση και βεβαίως δεν ήταν το πρόβλημα ε, σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα των εθελοντών για το ότι είχαμε μεγάλη έκταση στις πυρκαγιές. Ε, και να πω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει πολύ σοβαρές προσπάθειες και οι εθελοντές που προσφέρονται κάθε φορά για την κατάσβεση των πυρκαγιών είναι κάθε φορά και περισσότεροι και πιο οργανωμένοι. Θέλω όμως, και γι' αυτό πήρα το λόγο, να κάνω μια ειδική αναφορά στο παράδειγμα που είχαμε εμείς στην Ελλάδα το 2004 στην διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που νομίζουμε ότι η διοργάνωση αυτή κατεγράφει ε, ιστορικά ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Θυμάμαι τότε στην Ελλάδα ότι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και το προηγούμενο διάστημα όταν είχαμε την εκπαίδευσή τους και είχαν κάνει δικό τους κτήμα, ένιωσαν δική τους υπόθεση τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχαν φορούσαν όλοι τότε θυμάμαι τα μπλουζάκια τους, είχαν τον εξοπλισμό τους και πραγματικά η, εικόνα εκείνη έχει μείνει χαραγμένη σε όλους μας ως μια από τις καλύτερες εικόνες ε, της σύγχρονης Ελλάδας. Το λέω αυτό γιατί αν σε κάτι κάνουμε αυτοκριτική μας στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι στη συνέχεια δεν αξιοποιήσαμε όσο θα θέλαμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε όλο αυτό το μεγαλείο εκείνης περίοδου και δυστυχώς στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε με την ίδια ένταση την εθελοντική προσφορά των Ελλήνων. Το λέω αυτό για να καταλήξω στο εξής. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ονομάσαμε το 2011 έτος εθελοντισμού ή ενδεχομένως να έχουμε και κάποια παραπλήσια ονομασία όπως λέει ο κύριος Σκούρια. Εγώ νομίζω ότι ο τίτλος πάντως ε, είναι απολύτως κατανοητός από τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως το 2011 να αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια στις δράσεις που θα κάνουν οι οργανώσεις και όλοι οι εκπρόσωποι φορέων το 2011 και ό,τι προσπάθεια αφιερώσουμε στο 2011 να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, να μην έχουμε μια ενθουσιώδη προσπάθεια το 2011 και στη συνέχεια να μην έχουμε αντίστοιχη πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Τώρα κλείνω ο κατάλογος ομιλητών. Έναν ακόμα έχω στον κατάλογο αυτό. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι με είχατε δει πρόεδρε όταν ζήτησα το λόγο. Λοιπόν, θέλω να επιμείνω σε κάτι που θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γλωσσικό λάθος η χρήση του όρου βολοντεριά. Το θέμα δεν είναι νομικό, είναι το θέμα πώς μεταφράζεται στα γαλλικά. Οι Γάλλοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και ξέρουν πολύ καλά πώς πρέπει να μεταφράζουμε έναν όρο. Λοιπόν, όταν το volunteer το μεταφράζουμε ως βολονταριά στα γαλλικά, δεν συμπεριλαμβάνουμε την έννοια της κοινωνικής εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να αλλάξει αυτό. Κύριε Σιγητά, δεν σας ευχαρίστησα, συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Και θέλω να επιμείνω στο ζήτημα ε, του τι πρέπει να προσέξουμε κάθε φορά που μιλάμε για μια βάση δεδομένων. Είμαι στην Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη, όπου μας απασχολεί πάρα πολύ το εντό αγωγικών φακέλωμα. Δηλαδή το ότι διατηρούμε δεδομένα και στοιχεία όλο και περισσότερο. Όταν φτιάχνουμε ένα αρχείο για μία ένωση, για ένα σύλλογο εκεί, μπορεί να εμφανιστούν διάφορες δραστηριότητες πολιτικές, εδεκαλιστικές, θρησκευτικέ των ατόμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την οργάνωση, σε αυτή την ένωση. Λοιπόν, πρέπει να επιμείνουμε στο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, κάποια στοιχεία προφύλαξης, προσοχής. Η κυρία Σβένσον, για παράδειγμα, μίλησε για το mainstreaming των δύο φύλων. Και εδώ. Και γι' αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τη διάσταση των δύο φύλων όταν πρόκειται για θελοντές. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να ξέρουμε ότι πάρα πολύ πρόθυμες είναι αλλά δυστυχώς, όπως κι αλλού, όσο ανεβαίνουμε στη... στις ευθύνε που έχει κάποιος, οι γυναίκες εξαφανίζονται. Έπειτα για την χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτή τη διάσταση των δύο φύλων στις αποφάσεις της. Τέλος. Για τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών οργανώσεων. Συγχρόνω βέβαια πρέπει να σα πω ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχουν οργανώσει που πράγματι δεν χρειάζονται λεφτά. Δεν ζητάνε εξάλλου, είτε μικρέ είτε μεγάλε. Αν όμω θέλουμε οι μικρέ οργανώσει. Αυτέ που βασίζονται μόνο στον εθελοντισμό, να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, και ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι διαδικασίες, είναι αναγκαίο να έχουμε ειδικά μέσα ώστε να βοηθούμε τις μικρές αυτές οργανώσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Τέλος, είναι δυνατόν να ετοιμάσει κανείς έκθεση για αυτό το θέμα χωρίς να θίγει και το θέμα των κοινοφελών υπηρεσιών. Στη Γαλλία βλέπετε έχουμε μιλήσει πολύ για τους δίκτες αναγνώρισης κοινοφελών υπηρεσιών και ποια είναι η θέση των εθελοντών μέσα σε αυτές. Και εδώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό το ζήτημα ακόμα και αν φύγετε και σε άλλους χώρους. Ευχαριστώ. Ωραία, είχα πει ότι θα έκλεινα τον κατάλογο. Η κυρία του όμω είχε ζητήσει το λόγο στο μεταξύ και βέβαια πρέπει να το δώσω. Ναι, ναι. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να πω ότι ανάμεσα στα 6, 12 εκατομμύρια έτσι κι αλλιώς τα χρήματα δεν θα είναι ποτέ ε, αρκετά για να προωθήσουμε το έργο των εθελοντών. Εδώ δεν λέμε όμως συγκεκριμένα στην έκθεση ποιος το οργανώνει. Μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξουν ε, προσφορές, κάποιοι θα κερδίσουν. Ίσως αυτή τη φορά για το έτος εθελοντισμού να μπορούσαμε να οργανώσουμε το διαγωνισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακριβώ αυτοί που θα κερδίσουν εθελοντέ. Να είναι μια θελοντική οργάνωση που θα το αναλάβει, που θα οργανώσει όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο έγγραφο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας όλους τώρα. Εκπρόσωπος, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τα όσα σχολιάσατε. Πρώτα απ' όλα. Βλέπω ότι τα δύο κοινοτικά όργανα βρίσκονται δίπλα-δίπλα, πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Άρα φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία. Στο Συμβούλιο με ξέπληξε η ομοφωνία που έδειξε το Συμβούλιο για την απόφαση, αφού βέβαια συζήτησα διάφορα πρακτικά ζητήματα, εννοείται, αλλά πραγματικά υπάρχει ομοφωνία. Και από αυτά που άκουσα εδώ, ακόμα και να έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις, τίποτα δεν υπάρχει που να με εκπλήσει. Ξεκινάω από την ιδέα για μια βάση δεδομένων. Έχουμε επιφυλάξεις. Σκεφτείτε μια βάση δεδομένων για τον εθελοντισμό που να περιλαμβάνει όλου του εθελοντέ μετά από αυτά που ακούσαμε από την κυρία Τζάκια, την ευαισθησία των δεδομένων. Πώ θα τα διαχειριστεί κανεί αυτά. Αυτά αλλάζουν κάθε μέρα. Η Επιτροπή ποτέ δεν θα καταφέρει να τα διαχειριστεί. Μίλησε με την κοινωνία των πολιτών, κατά πόσο εκείνη μπορεί να ενημερώνει τα δεδομένα αυτά. Όχι, δεν είναι έτοιμη. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να σκεφτούμε μια πύλη, ένα πορτάλι, πόρταλ, που να μπορούμε να στείλουμε σε διάφορα links όλα όσα γίνονται με τον εθελοντισμό είτε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είτε στις κυβερνήσεις και για να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας Μακίν, η οποία μετέφερε σχόλια για ερωτήσεις άλλη συναδέρφου, η ενημέρωση των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή, με τη βοήθεια όμως της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο πόρταλ η Επιτροπή. Δεύτερη παρατηρήσή μου για την συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή πρότεινε να πάμε μέχρι το 80% για διάφορους καλούς λόγους. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα να πάμε μέχρι το 80%. Τρίτη παρατήρηση που θέλω να σας κάνω. Πρόκειται για τον τίτλο οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου είπαν ότι ο θελοντισμός δεν είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας κομψός τρόπος στήριξης, νομικής στήριξης στον εθελοντισμό και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την ηθαγένεια, την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ε, δεν είχαμε συζητήσεις με την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βλέπουμε ότι είναι ένας καλός τρόπος για να λυθεί αυτό το νομικό ζήτημα. Όμως εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι κάθε φορά που θα μιλάμε για αυτό το θέμα θα χρησιμοποιούμε τον όρο συν. Στην ανακοίνωση φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τον σύντομο τίτλο και εννοείται ότι στα γαλλικά θα κάνουμε διαφοροποίηση όπως μας ζητάνε οι γαλλόφωνοι. Ας προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε για τον νομικό όρο, γιατί τον χρειάζονται οι νομικοί, αλλά κάθε φορά που θα το μεταφέρουμε στο κοινό προς τα έξω, θα συνοηθούμε μεταξύ μας τι θα κάνουμε. Για τον προπολογισμό. εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πρόταση, αλλά αυτή η πρόταση είναι το ελάχιστο το ελάχιστο προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε το έτος αυτό. Αλλά όχι για να χρηματοδοτήσουμε δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, δεν είναι με τα 6 εκατομμύρια που θα το κάνουμε. Επιπλέον προπολογισμό χρειάζεται. Και φυσικά η Κομισιόν δεν έχει καμία αντίρρηση. Όμως το Κοινοβούλιο είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί το περιθώριο λιγμών του. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη συνέχεια, να καταλήξουν δηλαδή στη χρηματοδότηση. Ό,τι αποφασιστεί, η Κομισιόν θα το υποστηρίξει και θα το εφαρμόσει. Ευχαριστούμε. Ωραίες οι απαντήσεις σας. Τέλος, τελευταία σχόλια. Τελικά σχόλια. Ο κύριος Σκούρια. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής γιατί νομίζω ότι αποσαφηνίσαμε κάποια ζητήματα. Όσον αφορά το όνομα τώρα, αυτά που μόλις ε, μας είπε και ο Βανέσσα νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτό που είχε, το, το πρόβλημα που είχε προκύψει ήταν καθαρά νομικό θέμα ε, και νομίζω ότι με τη λύση αυτή μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να ονομάσουμε για όλους ε, το έτος αυτό Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και να βάλουμε έναν υπότιτλο που θα ε, λύνει το νομικό ζήτημα έτσι ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Επίσης, μου ετέθη το ερώτημα εάν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Πρέπει να σας πω ότι ε, το χρονοδιάγραμμα είναι ε, συγκεκριμένο. Ήδη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην τελική έγκριση του κειμένου. Ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι την 23η ε, Νοεμβρίου έχει συγκληθεί ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα στην Ολομέλεια πάντα του Νοεμβρίου ε, και έτσι ώστε να υποβάλουμε τον πλήρη φάκελο στο Συμβούλιο εντός του χρονοδιαγράμματος. Όπως είπα και προηγουμένως κάποια στιγμή, είναι γεγονός ότι είναι πολύ ζορισμένο το χρονοδιάγραμμα. Κινηθήκαμε με πάρα πολύ ταχύτητα. Ε, σας είπα και πριν ότι έχετε ακόμα την ε, δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίες, αλλά ήθελα να πω επίσης αφενός ε, ότι όπως αναφέρεται και στην τροπολογία 6, ε, έχουμε ήδη σκεφτεί το να ε, εργαστούμε προς την δημιουργία ενός ε, web portal, μιας πύλης διαδικτυακής. Βεβαίως έχουμε επίσης προβλέψει συνεργασία με τους εθνικούς φορείς, έναν κοινό συντονισμό των δράσεων, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα το ζήτημα της συγχρηματοδότησης παραδόξως σχεδιάστηκε για να βοηθηθούν ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν μικρές δομές και άρα λιγότερα χρήματα. Τελικά ε, τα χρήματα αυτά κινδυνεύουν ε, ε, να οδηγηθούν προς τα πιο μεγάλα δίκτυα, προς τις πιο μεγάλες οργανώσεις. Αυτό μας δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Επαναλαμβάνω πάντως ότι και βάσει όσων μας είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ευελπιστούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα αυξηθεί. Και επομένως τότε μπορούμε να επανέλθουμε στη χρηματοδότηση του 80%. Να ολοκληρώσω, γιατί βιαζόμαστε να μην μας εγκαταλείψουν και οι διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, προλάβουμε να τα πούμε όλα πριν. Να κάνω και μία πολιτική θεώρηση, δηλαδή πιστεύω ότι και το 2010, κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έτους, που μπορούμε τεχνικά να προετοιμάσουμε τις δραστηριότητες, αλλά όχι μόνον αυτό. Πιστεύω ότι ήδη από το 2010 θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την τροχιά που θα είναι προετοιμασία του 2011 αλλά και που θα θέσει τις βάσεις μιας καλύτερης πολιτικής και κοινωνικής προσέγγισης του εθελοντισμού και αυτό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί Θέλουμε να αποφύγουμε ε, να τελειώσει το ευρωπαϊκό έτος το 2011 και μετά να μην ξαναμιλήσει κανείς για τον εθελοντισμό. Το 12, το 13 θέλουμε ε, να εξακολουθούμε να συζητούμε για τον εθελοντισμό. Θέλουμε να έχει προχωρήσει το ζήτημα ε, του εθελοντισμού και επομένως να μην έχουμε μονάχα ένα πυροτέχνημα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους αλλά να έχουμε ένα ακόμα λιθάρι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Να έχουμε δηλαδή δομέ τι οποίε θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου ε, που έθεσαν τα ερωτήματα. Ευχαριστώ όλου όσου ε, ε, συμμετέσχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην διαδικασία. Να ευχαριστήσω βεβαίω και την γραμματεία τη Επιτροπή μα που με βοήθησε πάρα πολύ, που δούλεψε, γιατί δουλέψαμε χέρι με χέρι με την Γραμματεία της Επιτροπής. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκούρια. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, λοιπόν. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 5η 12 Νοεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι. 5η 12 Νοεμβρίου λοιπόν στις 12 ακριβώς. Μετά θα έχουμε την έκτακτη συνεδρία του Στρασβούργου 23 Νοεμβρίου στις 9, έτσι ώστε να ε, συζητήσουμε, να ψηφίσουμε την... Ναι, 9 λέτε, ναι, 9 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Είναι στριμωγμένο το χρονοδιάγραμμα. Επομένως, ε, γι' αυτό να σας ζητήσω, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και για μετάφραση, αν μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας στα αγγλικά ή στα γαλλικά, θα ήταν εξαιρετικό. Αν είναι δυνατόν θα ήταν εξαιρετικό, λέω. Να υποβάλλετε τις τροπολογίες. Σημείο 9. Στις 9 το πρωί συνεδρίασαν και κλεισμένων των θυρών οι συντονιστές να σας σταλούν ε, τα αποτελέσματα της συνεδρίας αυτής των συντονιστών. Προτείνω εκ των προτέρων να δεχτούμε τις αποφάσεις αυτές των συντονιστών. Συμφωνείτε, ναι. Σας ευχαριστώ. Σημείο 10. Διάφορα. Υπό τα διάφορα θέλει κάποιος ε, να ε, υποβάλει κάτι. Όχι. Τελευταίο σημείο. Η ημερομηνία της προσεχού συνεδριάσεως, όπως ε, σας είπα, θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση την ε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Θα έχουμε μονάχα ένα θέμα, ψηφοφορία επί της εκθέσεως ε, Μάρκος Κουρία. Η επόμενη τακτική συνέδρια της Επιτροπής θα λάβει χώρα την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.